Λοιπόν, συνάδελφοι, καταρχάς θέλω να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ε, συνεδρίαση του 2017, το δεύτερο ήμιση της ε, νομοθετικής μας θητείας και ακόμα και αν έχουμε μπει στο δεύτερο ήμιση του Ιανουαρίου, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο για το 2017 για όλους σας. Το πρώτο, τα πρώτα πέντε σημεία της ημερήσιας διάταξης αφορούν την εκλογή του Προεδρίου της Επιτροπής μας. Για την ώρα εγώ Προεδρεύω ως απερχόμενος πρόεδρος ε, του πρώτου ημίσεως της θητείας, πάνω κάτω δηλαδή ως προσωρινός πρόεδρος, απερχόμενος. Αυτή είναι η παράδοση του Κοινοβουλίου να προεδρεύει ο απερχόμενος πρόεδρος στην συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα. Επ' αυτή μου την ιδιότητα λοιπόν ε, κηρύσω την έναρξη της ε, συνεδρίασης ε, της ίντα. Τα πρώτα πέντε λοιπόν σημεία αφορούν την εκλογή του Προεδρείου και η σειρά της, ε, των εκλογών θα είναι καταρχάς η εκλογή του Προέδρου, μετά εκλογή πρώτου, δεύτερου, τρίτου και τέταρτου αντιπροέδρου. Με ενημέρωσαν ότι ορισμένοι ε, αναπληρωματικοί βουλευτές θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Και θα πρέπει να σας θυμίσω να έχετε όλοι σας ε, την κάρτα ψηφοφορία σας. Μήπως, μήπως χρειαστεί ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αν έχετε επιθυμία να αλλάξετε ή να ε, Δηλώστε κάποια υποψηφιότητα, παρακαλώ να ενημερώσετε την γραμματεία πριν να ξεκινήσουν οι εκλογές. Μάλιστα. Οπότε, καταρχάς θα πρέπει να εκλέξουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής. Χρειάζεται καταρχά να ελέγξουμε την απαρτία. Χρειαζόμαστε 11 μέλη ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις εκλογέ. και σαφώς είστε εδώ περισσότεροι από 11 παρόντες. 27 για την ακρίβεια. Για να εκλεγεί ο εισερχόμενο πρόεδρος χρειάζεται να γίνει να υποβληθεί μια υποψηφιότητα από μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον από τρία μέλη της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ. Οι υποψήφοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν την δήλωση οικονομικών συμφερόντων τους, να την έχουν υποβάλει. Ε, έχει ζητηθεί ο λόγος από τους σοσιαλιστές. Μάλιστα, εξ ονόματος της ομάδας μου προτείνω τον κύριο Λάγκε ως πρόεδρο της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. There's no further nomination. Δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος. Και εγώ δέχομαι την ε, υποψηφιότητα και επίσης έχω υποβάλει την δήλωση οικονομικών μου συμφερέοντων. Δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Οπότε, σύμφωνα με το άρθρο 208, έχουμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε διαβοής. Thanks a lot for your support. Σας, σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας και βεβαίως θα συνεχίσω την προσπάθειά μου να είμαι πρόεδρος όλων των βουλευτών αυτής της Επιτροπής και να αντιπροσωπεύω όλα τα μέλη καθώς και να αγωνίζομαι για τα δικαιώματα αυτής της Επιτροπής, ώστε στο μέλλον να έχουμε καλές νομοθετικές ε, πράξεις και καλές εμπορικές συμφωνίες. Προς... Ε, θα κάνω λοιπόν ό,τι περνά από το χέρι μου. Σας ευχαριστώ όλους. Και τώρα προχωράμε στην εκλογή των αντιπροέδρων. Και εδώ έχουμε ε, κανόνες ε, στο άρθρο 208 που διέπουν την εκλογή των αντιπρόεδρων και να σα θυμίσω ότι σε αυτό το άρθρο 208 περιλαμβάνεται ο σεβασμός της ε, αρχής της γεωγραφικής προέλευσης και της εθνικότητας, άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι άλλος Γερμανός υποψήφιος. Πρώτος αντιπρόεδρος λοιπόν ζητάω υποψηφιότητες και δίνω το λόγο στον, στον συντονιστή του ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. και προτείνω τον Γιώργο Βίνκλερ, εξ του ΕΛΚ, που έκανε πολύ καλή δουλειά τα τελευταία δυόμιση χρόνια στην ίδια θέση. Είχα προχωρήσει λίγο παρακάτω στην ατζέντα. Ε, έκανα λάθος. Την κυρία Σαΐφη ήθελα να προτείνω για πρώτη αντιπροέδρο, που επίσης έκανε πολύ καλή δουλειά τα δύο προηγούμενα χρόνια. Ε, ζητώ συγγνώμη κυρία Σαΐφη. Δέχεστε την υποψηφιότητα κυρία Σαΐφη, μάλιστα. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες, όχι. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε διαβοήση. Madam Saifi, please join me here. Μπορείτε, μπορείτε να έρθετε στο Προεδρείο, κυρία Σαΐφη. Okay, now we are switching to the election. Τώρα θα ψηφίσουμε για τον δεύτερο αντιπρόεδρο. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Χάουταλα των Πρασίνων για να υποβάλει την υποψηφιότητά τους. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια σε εσά και στην κυρία Σαΐφη για την εκλογή σας. Εγώ θέλω να προτείνω τον Γιάννη Ζαντόβ για δεύτερο αντιπρόεδρο. Δυστυχώς δεν είναι παρόν. Thanks uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζαντό έχει δεχτεί την υποψηφιότητά του γραπτός. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι? Όχι. Διαβοής λοιπόν ψηφίζουμε. Ωραία λοιπόν, εξελέγει ο κύριος Ζαντό δεύτερος αντιπρόεδρος. Συγχαρτήρια. Προχωράμε στην εκλογή του τρίτου αντιπροέθρου. υποψηφιότητε, δίνω το λόγο στον, στον συντονιστή του ΕΛΚΑ. Μάλιστα. Ε, τώρα θέλω να προτείνω τον σωστό άνθρωπο για τη σωστή θέση και άρα τον Ιούλιο Βίνκλερ για τη θέση του τρίτου αντιπροέδρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ιούλιος Βίνκλερ, λοιπόν. Δέχεστε Κύριε Βίνκλερ, μάλιστα, ευχαριστώ. Υπάρχει άλλος υποψήφιος? Όχι. Προτείνω να τον εκλέξουμε δια Mr. Winkler, please. Ah, και τώρα, τε, εκλογή του τέταρτου αντιπροέδρου, υποψήφι κύριος Κάμπερ. Ευχαριστώ πρόεδρε, συγχαρητήρια για τη θριαμβ... θριαμβώδη σας επιστροφή και θέλω να προτείνω το συνάδελφο Ζαρεντό που ήδη έχει υπηρετήσει και αγαπά τη ροκ μουσική Θέλω λοιπόν να τον προτείνω ως υποψήφιο για την τέταρτη αντιπροεδρία. Ευχαριστούμε. Δέχεστε την υποψηφιότητα. Ωραία, ευχαριστώ. Άλλοι υποψήφοι υπάρχουν. Όχι. Τότε μπορούμε να ψηφίσουμε διαβοής. Ωραία, εκλέγεστε ως τέταρτος αντιπρόεδρος λοιπόν. Παρακαλώ, ελάτε εδώ στο Προεδρείο κοντά μας. So, the Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι εκλογές για το Προεδρείο και μπορούμε να περάσουμε στην ε, κανονική μας τακτική ημερήσια διάταξη. Και πάλι να σας ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξή σας προς το Προεδρείο που είναι το ίδιο που είχαμε και στο πρώτο ήμιση της ε, θητείας μας. Νομίζω ότι τα πήγαμε καλά. και ότι εργαστήκαμε προς το συμφέρον της Επιτροπής μας. Τώρα, έχουμε σχέδιο ημερήσια διάταξη για το υπόλοιπο τη συνεδρίασής μας. Είμαστε στο σημείο 6 αυτής, δηλαδή την έγκριση της ιδείας. Εάν δεν έχετε αντιρρήσεις, προτείνω λοιπόν να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Εγκρίνεται. Σημείο 7. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων, διαφόρων συνεδριάσεων μάλιστα, του, των περασμένων μηνών. Συνηθίζουμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά, να τα θεωρούμε μάλλον εγκεκριμένα, εφόσον δεν έχουμε λάβει σχόλια μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Και θα πράξουμε ομοίως. Παίρναμε τώρα στο σημείο 8, τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Η μερίστη διάταξη, όπως θα δείτε, είναι γεμάτη. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα προς συζήτηση. Ήδη σήμερα θα, θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με ε, τον Ομόδιο Επίτροπο για την Συμφωνία ΣΕΤΑ. Αύριο θα ψηφίσουμε για τη συμφωνία αυτή. Μετά θα συζητήσουμε τις προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου. Θα ε, συζητηθεί επίσης η διαδικασια αντι anti-dumping, πολυμερείς διαπραγματεύσεις δικαστήριο για, τις επενδυτικές, ε, για επενδυτικά θέματα και πολλά πολλά άλλα. Βλέπετε λοιπόν πως έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Γι' αυτό λοιπόν λίγες θα είναι οι ανακοινώσει μου. Πρώτα, για την ε, συνέχεια της ε, εντολής του κ. Σεβέντο, Γενικού Γραμματέα του ΠΟΕΠ, ζήτησε, και ε, ζήτησε εντολή. Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή υποψηφιότητων ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2016. Δεν υποβλήθηκαν άλλε υποψηφιότητε. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Άσε θα παραμείνει Γενικό Γραμματέα του ΠΟΕ. Μετά, να σα ενημερώσω επίση ότι οι διαπραγματεύσει για τη συμφωνία TTIP δεν έχουν προχωρήσει προς το παρόν, όμως και οι δύο εταίροι μέχρι το τέλος της θητείας του Προέδρου Ομπάμα συνέταξαν ένα έγγραφο απολογισμού αν θέλετε το οποίο δημοσιοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου και στο έγγραφο αυτό αναφέρονται οι δυσκολίες που συναντήσαν οι διαπραγματεύσεις και τα διάφορα επιμέρους σημεία έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τα μέχρι τώρα επιτεύγματα. Τι έχουμε καταφέρει και τι όχι στην ε, συμφωνία TTIP. Επίσης υπάρχει μια νέα μελέτη για τους ενδεχόμενους ε, εμπορικούς φραγμούς. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη από τους ε, συνεργάτες μας και αξίζει να τη διαβάσετε. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι την Πέμπτη θα γίνει η πρώτης θα, μάλλον ψηφίστηκε σε πρώτη ανάγνωση η συμφωνία για, την, ε, για τα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα της Λευκορωσίας. Αυτά λοιπόν από μένα. Τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα την Επίτροπο κυρία Μάλιμστρομ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία ΣΕΤΑ, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Οι συζητήσεις για την συμφωνία αυτή ήταν πάρα πολύ έντονες και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σταθήκαμε πολύ κοντά σε όλα τα στάδια. Δουλέψαμε εντατικότατα τους τελευταίους 12 μήνες έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να σας ενημερώσω πως εννέα φορές στην Επιτροπή Ίντα είχαμε ε, ανταλλαγή απόψεων με διάφορους ε, φορείς. Είχαμε τρία εργαστήρια για την ΣΕΤΑ που αφορούσαν τις διαφορετικές πτυχές της συμφωνίας και δύο φορές άλλη μία αντιπροσωπεία στον Καναδά από την Επιτροπή μας, η οποία συναντήθηκε για να συζητήσει επιμέρους λεπτομέρειες με τους ε, εταίρους του Καναδά. Επίσης, ε, διεξήχθησαν πολλές συζητήσεις με τα εθνικά κοινοβούλια Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολλά κράτη-μέλη για πρώτη φορά είχαν τη δυνατότητα να μας εκθέσουν τις δικές τους απόψεις. Και επίσης χρησιμοποίησαμε και τις ε, νομικές μας υπηρεσίες για να εξετάσουμε ε, το θέμα του επενδυτικού δικαστηρίου και να συζητήσουμε τις επιμέρους ε, πτυχές ερμηνείας της νομοθεσίας σχετικά. Όλες λοιπόν αυτές οι εργασίες οδήγησαν βήμα προς βήμα στην σημερινή μας ε, κατάληξη. Έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά στο τέλος. Να σας υπενθυμίσω ότι καταφέραμε να αλλάξουμε το ε, παλιό σύστημα που είχε προταθεί, το ISDS, το σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτή και κράτους και να το μεταμορφώσουμε σε ένα επενδυτικό δικαστήριο. Εξετάσαμε λοιπόν όλες τις νομικές πτυχές έτσι ώστε να φροντίσουμε να υπάρχει νομική προστασία για όλους τους ε, φορείς, να υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιώματα και συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις για τους εργοδότες, για τους εργαζόμενους, να γίνονται σεβαστοί τα δικαιώματα των εργαζομένων κτλ. Μετά λοιπόν από αυτές τις εντατικότατες συζητήσεις και μετά τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων, αγαπητές κυρίες και κύριοι, καταλήξαμε σε τρία θέματα στα οποία εστιάσαμε. Καταρχάς, οι μικτές επιτροπές, η μικτή επιτροπή για την ε, Συμφωνία ΣΕΤΑ, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την επιτροπή, ποια θα είναι η σύστασή της. Εδώ να σας πω ότι όπως και στις άλλες μικτές επιτροπές έχουμε το δικαίωμα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ενημέρωση. Έχουμε το δικαίωμα της ε, συμμετοχής σε αυτή την μικτή επιτροπή. Ωστόσο, σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στην συνεργασία μας και θα ήθελα να ξέρετε ότι και ο κύριο Μπροκ και εγώ βρισκόμαστε σε στενές διαπραγματεύσεις με τους υπόλοιπους έτσι ώστε να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στείλαμε λοιπόν μαζί με τον κύριο Μπρόκ μια επιστολή στο Συμβούλιο όπου αναφέρεται ακριβώς αυτή η επιθυμία μας, ότι δηλαδή θέλουμε ε, η μεικτή αυτή επιτροπή να ε, βελτιωθεί και αυτό να ε, υπάρχει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και να υπάρχει αγκυροβολημένο και στη συμφωνία έτσι ώστε να βελτιωθούν οι δημοκρατικές δομές Αυτά λοιπόν ως προς τη συνεργασία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Μετά, ο δεύτερος τομέας στον οποίο σταθήκαμε είχε να κάνει με την δήλωση υπαριθμών 36 για την περαιτέρω εξέλιξη δηλαδή του επενδυτικού αυτού δικαστηρίου. Και σταθήκαμε μάλιστα στο θέμα της επιλογής των δικαστών. Εδώ, κυρίες και κύριοι, θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μοντέλο με εκείνο του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εδώ θα έχουμε το δικαίωμα συμμετοχής και τρίτο θέμα στο οποίο σταθήκαμε είναι το τι γίνεται σε περίπτωση παραβίασης των εργατικών δικαιωμάτων. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις ασφαλιστικές ε, δικλείδες εκεί και πώς μπορούμε να συντάξουμε ένα σχέδιο δράσης, ένα χάρτη πορείας. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας λοιπόν. Αυτοί λοιπόν ήταν οι τρεις τομείς στους οποίους σταθήκαμε κατά τη διάρκεια των ε, συζητήσεων και διαπραγματεύσεών μας και θα συνεχίσει αυτή η συζήτηση σήμερα με την παρουσία της κυρίας Επιτρόπου, στην οποία θα δώσω ευθύ αμέσω το λόγο. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Λάγκε, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλό απόγευμα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με την ευκαιρία επίσης να σας συγχαρώ κύριε Λάγκε για την επανεκλογή σας ως, στη θέση του Πρόεδρου της Επιτροπής. Προσβλέπω θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με το ίδιο επικοδομητικό πνεύμα που είχαμε στη συνεργασία μας μέχρι σήμερα. Είναι κοινότοπο να πω ότι οι εποχές είναι περίπλοκες, δύσκολες, αβέβαιες. Φαίνεται ότι η νέα ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών θα ακολουθήσει μια νέα άλλη προσέγγιση στο διεθνές εμπόριο, στη θέση της διεθνής σκηνή και αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που πιστεύουμε ότι είναι εφικτό να καταλήγουμε σε διαφανείς, ε, ε, υποφελείς προς όλους τους πολίτες εμπορικές συμφωνίες, θα πρέπει να εντείνουμε τις συμμαχίες μας με εκείνους που σκέφτονται με τρόπο παρόμοιο με εμάς, για να αποδείξουμε ότι αυτές οι συμφωνίες λειτουργούν. Και ο καλύτερος σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια δεν είναι άλλος παρά ο Καναδάς, που είναι ε, μια χώρα με την οποία έχουμε εμπορικές συναλλαγές της, της τάξης του 3 εκατομμυρίου ευρώ και άμεσες επενδύσεις ε, πολλών δισεκατομμυρίων. Είναι ένας ε, εταιρός με τον ε, οποίο συμφωνούμε στα ζητήματα της, του κράτους δικαίου, της συμμετοχής των πολιτών, της διαφάνειας, της ασφαλιστικέ δικλείδε που πρέπει να υπάρχουν στι δημόσιε προμήθειε, στο εργατικό δίκαιο, αλλά επίση και σε άλλα ζητήματα όπω το θέμα τη κλιματική αλλαγή. Ο Καναδά συμφωνεί με εμά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η ε, εμπορικές συμφωνίες μπορούν να ε, καταπολεμήσουν την ενεργεία, μπορούν να δώσουν ε, νέες ευκαιρίες στους πολίτες μας και με αυτόν τον τρόπο να μας βοηθήσουν να δώσουν εμείς την κατεύθυνση που θα θέλαμε στην παγκοσμιοποίηση παρά να την ακολουθούμε. Είχε Είχα την ευκαιρία να αναπτύξω και ενώπιον σας στο παρελθόν τις αρετές της σχέσης μας με τον Καναδά. Όπως γνωρίζετε, ότι το, το γεγονό ότι θα καταργηθούν οι δασμοί από την πρώτη ημέρα σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρει να εξοικονομήσει 500 εκατομμύρια ε, ευρώ ετησίω. Αυτό θα ε, βοηθήσει κυρίω τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα προωθήσουμε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα τα οποία ε, παράγονται στον Καναδά, ποιότητα σε φάμιλες με εκείνα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εξαγωγές του ε, Καναδά ανέρχονται στα 11,5 δισεκατομμύρια ε, το χρόνο. Ε, οι τομείς της οικονομίας στις οποίες δραστηριοποιούνται, στις οποίες θα μπορούσαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να δραστηριοποιηθούμε, καλύπτουν την πληροφορική, τα σιδηροδρόμους και άλλους, την αυτιλία. Είναι τομείς αυτού στου οποίου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσει θα μπορέσουν να επενδύσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια, δημιουργώντα θέσει εργασία. εργασίας. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστέ και επιχειρηματίε θα μπορέσουν να παράσχουν συμπληρωματικέ υπηρεσίε σε καναδικέ εταιρείε. Έχουμε σημαντικέ ασφαλιστικέ δικλείδε σε αυτή τη ε, συμφωνία για τον, τη γεωργία όπου θα διατηρηθούν οι δασμοί για κρίσιμα προϊόντα όπως τα γαλακτοκομικά ή τα πουλερικά. Έχουμε επίση ακολουθήσει την προσέγγιση τη δημιουργία ενό δικαστηρίου για την επίλυση των επενδυτικών διαφορών. Ε, και γνωρίζω ότι πολλά από τα μέλη τη Επιτροπή έχουν υποστηρίξει αυτή την προσέγγιση. Έχουμε πολλέ φορέ ανταλλάξει απόψει σε αυτό το θέμα και με έχετε βοηθήσει να καταλήξω στην λύση που τελικά επελέγει. Ε, που είναι πολύ καλύτερη από το προηγούμενο σύστημα, το ISDS, γιατί διασφαλίζει το δικαίωμα της κυβέρνησης να ε, υιοθετεί το ρυθμιστικό πλαίσιο που επιθυμεί. Ε, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από κατακτισμένους δικαστές και θα διασφαλίζεται το δικαίωμα εφησυβολής της απόφασης. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, γιατί εμείς θα θέλαμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε πολυμερές επίπεδο διεθνώς, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα διεθνές τέτοιου τύπου δικαστήριο. Συζητήθηκε το θέμα μας με 27 υπουργού οικονομικών στον Ταβός και διαπιστώνω ότι πολλές χώρες στον κόσμο θέλουν να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο σύστημα. Μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες αν το επιθυμείτε. Με τη συμφωνία αυτή διασφαλίζεται επίσης ο δημόσιος χαρακτήρας των υπηρεσιών που επιθυμούν να διατηρήσουν δημόσιες οι Ευρωπαίοι, όπω το τομέα τη παιδεία, τη υγείας, είναι κάτι το οποίο επιθυμούν και οι Καναδοί. Ε, οι τοπικές ε, και περιφερειακές ε, αρχές και κυβερνήσεις να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τη δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών τους. Δεν υπάρχει υποχρέωση ιδιωτικοποίηση κανένα τομέα, ούτε η υποχρέωση να μην επανεθνικοποιηθεί κάποιο τομέα που ειδικοποιήθηκε. Με αυτόν τον τρόπο η ΣΥΤΑ επίσης προστατεύει και μια σειρά δικαιωμάτων, των περιβαλλοντικών, των εργατικών δικαιωμάτων, της προστασίας της διαφορετικότητας. Πολλά μέλη της Επιτροπής μας υπέβαλαν ερωτήματα, το ίδιο και πολλά μέλη της κοινωνίας και πολυπολίτες. Είναι λογικό, είναι φυσικό να λαμβάνετε τις ερωτήσεις των πολιτών που εκπροσωπείτε και να τις μεταφέρετε στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν να διευκρινίσω τρία θέματα που συζητήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Πρώτα απ' όλα ο Πρόεδρος ήδη αναφέρθηκε στο ζήτημα της μεικτής Επιτροπής ΣΥΤΑ, ποιο θα είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι αρμοδιότητές του. Και θα ήθελα να είμαι ξεκάθαρη. Τίποτα στην ΣΥΤΑ δεν επιτρέπει σε αυτήν την Μικτή Επιτροπή να παρακάμψει τις ε, πρόνοιες ε, της των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οποίο σημαίνει ότι αυτή η Επιτροπή, η Μικτή Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα μόνο μερό να τροποποιεί την ΣΥΤΑ. Οποιαδήποτε τροποποίηση της ΣΥΤΑ θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια δικασία που ακολουθήθηκε για την κύρωση της ΣΥΤΑ, δηλαδή πρόταση της Επιτροπής, απόφαση του ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το οποίο με λίγα λόγια σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση το κείμενο της ΣΥΤΑ δεν πρόκειται να αλλάξει χωρίς τη δικιά σύμφωνη γνώμη. Ε, υπάρχει η δυνατότητα ε, τροποποίησης παρατημάτων, αλλά και αυτή είναι περιορισμένη αυστηρά. Δεν μπορούν να τροποποιηθούν κρίσιμα παραρτήματα και πρωτόκολλα, όπως για παράδειγμα εκείνο που διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών. Μόνο όταν η συμφωνία ρητά επιτρέπει στην Μικτή Επιτροπή να κάνει τροποποιήσεις, μόνο τότε αυτό επιτρέπεται και θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη και της Ευρωπαϊκής Πλευράς, της της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πλευράς του Καναδά. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώ δεν πρόκειται να προχωρήσει σε ένα τέτοιο βήμα αν δεν έχει λάβει την σχετική εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Όταν ε, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση απαιτεί αλλαγή του ευρωπαϊκού δικαίου στι σπάνιες αυτέ περιπτώσει, περιπτώσεις, προφανώς θα σεβαστούμε τι δικέ μα εσωτερικέ διαδικασίε και δεν πρόκειται να δώσουμε τέτοια συνένεση στην Ιχτή Επιτροπή, εάν δεν τελειώσει αυτή η διαδικασία. Πολλοί έχουν εκφράσει φόβου για τις ζητήματα της, διατροφη... των τροφίμων, μάλλον και τη προστασία τη υγεία του καταναλωτή. Δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο. Εμεί, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τι συνήθει μα διαδικασίε, θα λαμβάνουμε και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τι αποφάσει μα για την προστασία τη ασφάλεια του καταναλωτή ε, της ασφάλειας των τροφίμων. Αυτό δεν αλλάζει και δεν μπορεί να αλλάξει με αποφάσεις της ε, Μεκτής Επιτροπής ε, της ΣΥΤΑ. Είναι ένα θέμα στο οποίο δώσαμε μεγάλη έμφαση, το προσέξαμε πολύ και οι Καναδοί και εμείς, γιατί και οι δύο πλευρές θέλουν να διατηρήσουν το δικαίωμα των δημοσίων αρχών τους να υιοθετούν ρυθμιστικά κανονιστικά μέτρα. Ε, ε, ε, τέθει επίση το ζήτημα του εάν θα πρέπει να αναβληθεί η υιοθέτηση τη ΣΥΤΑ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των διαπραγματεύσεων για τις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό δεν, το πιστεύω, δεν πιστεύω ότι είναι απαραίτητο, γιατί οποιαδήποτε και αν είναι συμφωνία τελικά καταλήξουμε και το Συμβούλιο και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα τη σεβαστούν, θα σεβαστούν την ισορροπία που θα βρεθεί. Είναι κάτι για το οποίο μπορεί να σα δώσει διαβεβαιώσει και ο πρόεδρο σα που συμμετέχει όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ε, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να υλοποιήσουμε ως Επιτροπή τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την τρέχουσα διαθεσμική συμφωνία ενημερώνοντα πάντα και την Επιτροπή Εμπορίου του Κοινοβουλίου. Γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι για εσά αυτό, ε, ε έχοντα την εμπειρία τη συνεργασία τα τελευταία 6,5 χρόνια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό πάντοτε, οποτεδήποτε μου ζητούσατε πληροφορίε, ε, απαντούσα ε, λεπτομεριακά. Όπως, Όπω για παράδειγμα η αναλυτική απάντηση που έδωσα στην επιστολή που έλαβα τον κύριο Μόισερ, με τον οποίο ευχαριστώ με την ευκαιρία. Η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων είχε σχέση με αυτό το νέο σύστημα το δικαστικό, το Δικαστήριο Επενδυτικών Διαφορών. Ε, δημιουργείται, όπως γνωρίζετε, ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ένα εφετείο και ε, ρυθμίσεις όσον αφορά τη διοντολογία και τον ορισμό των δικαστών. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα, ελέγχει την υλοποίηση, την εφαρμογή αυτή τη συμφωνία. Όπω είπα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μεγάλο βαθμό έχει διαμορφώσει αυτό το σύστημα και σα ευγνωμονώ για αυτό. Γι' αυτό και είμαι σίγουρο ότι και στο μέλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητηθεί ουσιαστικά και ει βάθο ε, αυτά τα ζητήματα ε, πριν προχωρήσουμε, πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε, για παράδειγμα, αλλαγή στο κείμενο της συμφωνίας που μπορεί να χρειάζονται Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θα για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θα ακολουθηθούν οι συνήθειε διαδικασίε για την κύρωση συμφωνιών, δηλαδή θα περάσουν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω επίση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει στον ορισμό των δικαστών. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να προτείνει ω πρόεδρο του δικαστηρίου έναν δικαστικό εγνωσμένου κύρου, ίσω πιθανώ κάποιο πρώην μέλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ε, να προεδρεύσει μια ε, επιστροπή η οποία θα γνωμοδοτήσει για την επάρκεια των υπολείπων προτινόμενων δικαστών. Ε, έχουμε την εμπειρία και τη γνώση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Ο κύριος ε, Λάγκε μου απέστειλε σχετική επιστολή και η αναλυτική μου απάντηση βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας. Το, η τρίτη ομάδα ερωτημάτων έχει σχέση με την βιώσιμη ανάπτυξη, ένα πολύ σημαντικό θέμα ε, διεθνώς, αλλά εγώ θα το δω από την πλευρά της ΣΥΤΑ. Έχουμε μπροστά μας μια συμφωνία η οποία διατυπώνει ρητά ότι το εμπόριο και η ανάπτυξη πρέπει να γίνονται με τρόπο βιώσιμο που να σέβεται ε, τα εργατικά δικαιώματα με προβλέψει σε αυτή η συμφωνία, οι οποίε είναι και νομικά δεσμευτικέ και άρα μπορεί να λειτουργήσει ω μοντέλο για όλο τον υπόλοιπο ε, κόσμο. Ε, καταγράφεται η υποχρέωση, για παράδειγμα, ε, προώθησης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντο, όπως για παράδειγμα τη Συμφωνία των Παρισίων, ε, της τήρησης των κανόνων του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου, όσον αφορά τι συλλογικέ συμβάσει, την καταπολέμηση των διακρίσεων στους χώρου εργασία κτλ. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδά συμφώνησαν ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να υπονομεύσουν την τρέχουσα, το τρέχον επίπεδο προστασία του περιβάλλοντο και των εργατών. Ε, και έχουμε δημιουργήσει και έναν ειδικό μηχανισμό για την επίλυση διαφορών σε αυτούς τους τομείς. Ε, είναι προτεραιότητά μας να φροντίσουμε για την αποτελεσματική υλοποίηση και λειτουργία αυτού του μηχανισμού. Συναντήθηκα επίσης και με τον κύριο Σομπάνη, τον νέο ε, ε, Υπουργό Εμπορίου του Καναδά, ο οποίος συμφωνεί μαζί μα για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Βεβαίω όλα αυτά θα γίνουν και με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη κοινωνία των πολιτών που χρειάζεται να συνεχίσουμε να κάνουμε ένα διάλογο σε αυτό το θέμα. Για παράδειγμα πώ θα λειτουργήσει ο μηχανισμό ε, εφαρμογή και ο μηχανισμό επίλυση διαφορών. Θα αξιοποιήσουμε, όπως συμφωνήθηκε στην τελευταία σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά, ε, τη διαδικασία για τη, για τη συζήτηση ζητημάτων βιώσιμου εμπορίου. Στόχος μου είναι να ξεκινήσουμε άμεσα διάλογο με όλους τα ενδιαφερόμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά, ε, έτσι ώστε να γίνει αυτή η αξιολόγηση, αυτή η αναθεώρηση για την ε, βοήθεια, την παροχή βοήθειας για το εμπόριο. Ε, αξιοποιώντας και την εμπειρία άλλων κρατών και στόχος είναι να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, έτσι ώστε τα συμπεράσματα του ιστορικού μας διαλόγου να ε, ενσωματωθούν στις διαπραγματεύσεις που έχουμε με τον Καναδά. Αυτή η συζήτηση είναι και γενικότερη. Θα μπορούσε να μας δώσει κάποιες ιδέες για το πώς θα ε, λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της εμπορικής βοήθειας ε, και του βιώσιμου εμπορίου γενικότερα και πέρα από τον Καναδά. Συμπερασματικά, το, η συμφωνία την οποία συζητάτε σήμερα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και οικονομική αλλά επίσης και γεωπολιτική. Έχουμε έναν σύμμαχο με τον οποίο έχουμε την ίδια λογική, την ίδια φιλοσοφία, με τον οποίο θέλουμε να καταλήξουμε σε μια προσέγγιση που βοηθάει να σχηματίσουμε εμείς την παγκοσμιοποίηση που θέλουμε, προστατεύοντας το δημόσιο συμφέρον, είμαστε εμεί που επιθυμούμε ένα ανοιχτό εμπόριο που βασίζεται σε κανόνε ε, και που επιθυμούμε δημοκρατικές κοινωνίες. Η Καναδάς είναι ένας τέτοιος εταίρος. Δυστυχώς άλλοι εταίροι μας απομακρύνονται από αυτές τις αρχές και εμείς ε, ε, κύριε Πρόεδρε πρέπει να φροντίσουμε να αγωνιστούμε εναντίον αυτής της λογικής του, του προστατευτισμού και της απομάκρυνσης από αυτές τις αρχές. και νομίζω ότι η συνεργασία μας με τον Καναδά μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό. Πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς καθυστέρηση. Ελπίζω ότι θα δώσετε αύριο τη θετική σας ψήφο ως Επιτροπή στην Συμφωνία. Το ίδιο ευελπιστώ θα γίνει και στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ και άλλη μια φορά κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπε. Νομίζω πως ε, κατέστη σαφές από εσάς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει κάποιες πρόσθετες υποχρεώσεις στην επιλογή των δικαστών, για παράδειγμα, αλλά και για την ε, εφαρμογή ε, των, ε, της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για όλα αυτά. Θα σας συνοδεύουμε στο μέλλον σε αυτό το έργο. Έχετε την υποστήριξή μας. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές και μετά έχουν ε, ζητήσει το λόγο αρκετοί συνάδελφοι. Δεν θα δώσω συγκεκριμένο χρόνο ομιλίας, όμως ελπίζω να είστε σύντομοι και πάνω κάτω να μείνετε στα δύο λεπτά. Κύριε Παύριξ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε, για αυτό αυτές τις εξηγήσεις. Ήσασταν άμεση, περιεκτικότατη και σαφέστατη. Πράγματι, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια και εγώ θα αρχίσω από εκεί που σταματήσατε. Να υπενθυμίσω καταρχάς ότι εάν πράγματι επιθυμούμε να συνεχίσουμε στην προσπάθεια να βελτιωθούν οι σχέσει με του σημαντικού εταίρου όπω τον Καναδά. Αυτέ οι συμφωνίε είναι ο τρόπο με τον οποίο θα το πετύχουμε. Αν δεν δείξουμε την εμπιστοσύνη μα στου Καναδού, οι οποίοι να υπενθυμίσω ότι είναι ε, σαν και εμά, μοιάζουμε πάρα πολύ, τότε ποιον μπορούμε να εμπιστευτούμε. Μπορούμε να εμπιστευτούμε του ίδιου μα του εαυτού. Αυτό ω τροφή για σκέψη. Μετά, ω προ το περιεχόμενο, να επαναλάβω τις απαντήσεις που δόθησαν σε αυτές τις επιστολές προς την Επιτροπή και ε, να σας πω πως έχουν γίνει πολύ άριθμες συζητήσεις στο παρελθόν για αυτά τα θέματα. Καταρχάς, η Μικτή Επιτροπή είναι ένας πολύ καλός θεσμός, ο οποίος θα αποτρέψει τις ε, πιθανές διαφωνίες που ενδεχομένως προκύψουν. Ταυτόχρονα όμως θα διασφαλίζει την διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει αλλαγή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, εάν προκύψει τέτοιο θέμα. Όλα λοιπόν αυτά τα θέματα που ανησυχούν τους πολίτες μας σίγουρα θα ε, εξετάζονται από αυτήν τη μεικτή επιτροπή. Μετά, αυτό το διεθνές δικαστικό σύστημα, να πω πως πριν την ε, τωρινή συμφωνία είχαμε μια πάρα πολύ προηγουμένη πρόταση. Και το Κοινοβούλιο αλλά και οι πολίτες θα κληθούν να απαντήσουν στο ερώτημα τι ακριβώς ε, θέλουμε. Δεν τίθεται θέμα υπονόμευσης της ποιότητας των συμφερόντων, των κοινωνικών κεκτημένων, της υγείας ε, των πολιτών. Να πω μετά πως πιστεύω ότι όλα αυτά τα θέματα που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν έχουν λίγο πολύ απαντηθεί και πως είμαστε επιτέλους έτοιμοι να δώσουμε ένα τέλος σε αυτές τις ατέρμονες συζητήσεις και να ψηφίσουμε αύριο στην Επιτροπή μας. Η συζήτηση αυτή ήταν δημόσια και ελπίζω το Φεβρουάριο στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο, να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις και να δείξουμε ότι έχουμε πάρει την πρωτοβουλία για την βελτίωση των σχέσεων και για ένα, μια νέα σελίδα στις σχέσεις μας με τον Καναδά. Να ε, πω εδώ επίσης ότι ελπίζω να τηρήσουμε τις, υποχρεώσεις, τις ε, υποσχέσεις που έχουμε δώσει στους Καναδούς εταίρους μας αλλά και στους ίδιους μας τους εαυτούς. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μόησα. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω καταρχάς την ε, κυρία Επίτροπο για τις απαντήσεις στην επιστολή που στείλαμε και εμείς και εσείς κύριε Πρόεδρε. Οι απαντήσεις αυτές έφεραν σαφήνεια και έριξαν φως σε πολλά ζητήματα τα οποία θεωρούνταν ενδεχομένως εμπόδια για την τελική ψηφοφορία στη Συμφωνία ΣΥΤΑ. Νομίζω πως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που βλέπουμε επιτέλους φως στην άκρη του τούνελ. Βλέπουμε το τέλος της διαδικασίας, έχουμε κάποιες εγγυήσεις ότι το κείμενο, το κυρίως κείμενο δεν μπορεί να τροποποιηθεί από την Εμικτή Επιτροπή, αλλά μόνο ε, από τα ε, μέρη, ότι μπορεί να υπάρξει μόνο συμφωνία στο κείμενο. Ε, δεν αναφέρομαι στα παραρτήματα. Να πω επίσης ότι γιατί οποιαδήποτε απόφαση λάβει αυτή η μεικτή επιτροπή δεν θα βασίζεται σε παράκαμψη του ρόλου του Κυροβουλίου. Θα υπάρχει καταρχάς η εσωτερική κοινοτική διαδικασία, μετά θα γίνει μια αξιολόγηση από την Επιτροπή αυτής της διαδικασίας και θα υπάρχουν εγγυήσεις ότι η νομοθεσία μας δεν θα μπορεί να αποδυναμωθεί είτε έμεσα είτε άμεσα ε, εις βάρος μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες και μπορεί να δράσει σε αυτό το θέμα. Μετά, έχουμε επιτέλους μία εγγύηση όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μάλλον από το διπλό σύστημα ε, της νομοθεσίας μας, ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εφαρμογή νομοθεσίας. Δεν θα μας αναγκάσει δηλαδή η συμφωνία ΣΥΤΑ να αλλάξουμε την νομοθεσία μας. Ε, πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό το επίτευγμα και για το ότι θα διατηρήσουμε την κυριαρχία μας σε αυτό το θέμα. Μετά, ε, χαίρομαι πολύ για τις απαντήσεις που δώσατε σχετικά με την εκλογή των δικαστών. Η διαδικασία της οποίας θα είναι παρόμοια με εκείνη του, της εκλογής των δικαστών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και χαίρομαι πολύ για το ότι αναφέρεται πως θα γίνει μια δημόσια διαβούλευση έτσι να οδηγηθούμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σχετικά με τις κυρώσει και με την επίλυση ε, διαφορών. Τώρα, να πω ότι πιστεύω πως η ομάδα μου έχει προσπαθήσει πάρα πολύ να προωθήσει μια προοδευτική ατζέντα και για ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη και για όλους μας και για τη συμφωνία αυτή. Εμείς στηρίζουμε τη συμφωνία ΣΥΤΑ. Γι' αυτό λοιπόν αύριο στην ψηφοφορία θα ταχθώ υπέρ μια θετικής ψήφου, ε, αλλά όχι μόνο αύριο και στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Κάμπερ. Πρόεδρε, Επίτροπε, εγώ και η ΣΥΑΡ είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που η ΣΥΤΑ επιτέλους ε, πλησιάζει στο τέλος μετά από τόσες ε, ανώφελες καθυστερήσεις. Θα την υπερψηφίσουμε αύριο και στο Στρασβούργο. Πιστεύουμε πως φτάνει πια. Πολλοί στόχοι έχουν ξεκαθαριστεί και σας ευχαριστώ που το κάνατε αυτό. Ε, στην Κοινή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ για τη σκληρή δουλειά της DG Trade στην ε, πλευρά των διαπραγματεύσεων. ε, για κάτι πιο γενικό. Η ΣΥΤΑ δεν περιλαμβάνει ελεύθερη κυκλοφορία και δεν περιλαμβάνει ε, τέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάει για στρατηγική εταιρική σχέση που χρησιμοποίησε και ο Πρωθυπουργό μα την περασμένη εβδομάδα. Εσεί βλέπετε με κάποιο τρόπο αυτό να είναι καλό πρότυπο για μια μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου. Γιατί, όπω είπατε, είναι μια πολύ καλή σύγχρονη συμφωνία και με άλλα έθνη ίσω. Και Νομίζω πως ε, εφόσον θα πρέπει κάποια λύση να βρεθεί, θα μπορεί αυτό να είναι μια επιλογή. Ο Καναδάς έχει την ίδια βασίλισσα, είναι ε, ε, ακλόφωνος, έχει τους ίδιους κανόνες. Τι ίδιε νομοθεσίε έχουμε πολλά κοινά και επίση η οικονομία υπηρεσιών είναι ένα καλό παραλληλισμό. Έχετε τίποτα να μα πείτε κατά πόσο είναι ένα καλό τρόπο να προχωρήσουμε γενικότερα και ευρύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Και ευχαριστώ, ευχαριστώ την ε, Επίτροπο και την, το επιτελείο της για αυτό τον μαραθώνιο ε, της ε, ΣΕΤΑ που ελπίζω πως θα ολοκληρωθεί σύντομα. Με ικανοποίηση άκουσα ότι εσείς επιβεβαιώσατε τα προσεκτικά βήματα που κάναμε τα τελευταία 7 χρόνια. Πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να φτάσουμε όμως σε ένα καλό τελικό αποτέλεσμα. Επίσης είμαι ευγνώμων για τα όσα είπατε στην αρχή της δήλωσής σας για τις ε, δύσκολες ε, ε, περιόδους που περνάει ο κόσμος, η Ένωση αλλά και η Δηλαδή, δική μα σχέση. Πρέπει να είμαστε ε, ανοιχτοί, ειλικρινεί για το τι συμβαίνει, για το ανοιχτό χαρακτήρα των κοινωνιών μας, της οικονομίας μας και το ανοιχτό μυαλό μας. Κάτι που, για το οποίο πρέπει να αγωνιστούμε. Δεν χρειαζόμαστε εμπορική ατζέντα τύπου Τραμπ, αλλά περισσότερο τύπου Τριντό. Ε, μία που να καλύπτει και να αγκαλιάζει τις ευρωπαϊκές αξίες, τις ε, υψηλέ προδιαγραφές και θα εγγυάται το δικαίωμα να μπορούμε να νομοθετούμε. Μας επιτρέπει ώστε από κοινού να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε τους κανόνες των εμπορικών συστημάτων και να στηρίξουμε και το πολυμερές εμπορικό σύστημα το οποίο χρειάζεται υπεράσπιση. Δεν μπορούμε να βρούμε κανένα καλύτερο σύμμαχο, πιστεύω, από τους Καναδούς για να μοιραστούμε αυτές τις δύσκολες στιγμές, αλλά και να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε όσους θέλουν να προκαλέσουν και να αφισβητήσουν τις αρχές μας, τις αρχές που καθιστούν το επίπεδο διαβίωσής μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Καναδά. Για όσους ακόμα έχουν αμφιβολίες και που ε, αυτή τη στιγμή έρχονται με νέα ερωτήματα, είναι σαφές πως δεν έχουμε άλλο χρόνο να χάσουμε και ελπίζω πραγματικά ότι αύριο θα μπορέσουμε στην Επιτροπή μας και αργότερα στην Ολομέλεια να σχηματίσουμε μια ευρεία κεντρώα συμμαχία. Γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ήταν, και το λέω αυτό και στους Ιαλδημοκράτες, ήταν δουλειά πολλών ανθρώπων και πολύ θα ήθελα να επιτύχει και να μην δούμε διχασμούς. Ήταν ομαδική η προσπάθεια, ήταν δύσκολη, αλλά έχουμε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι με το τελικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Αν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, η βασική μου ανησυχία όταν μιλάμε για τη ΣΕΤΑ είναι η απειλή για τη δημοκρατία. Έχω ήδη διατυπώσει σχόλια ω προ αυτό το θέμα, αλλά έχω την εντύπωση πω έχουν μείνει νεκρό γράμμα και άρα επανέρχομαι δρυμύτερη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στόχο έχει να, να αντιπροσωπεύει του ευρωπαϊκού λαού και τα να στηρίζει τα συμφέροντα των συμπολιτών μα. Πρέπει να ενεργούμε έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα αυτά σε θέματα ασφάλεια, διατροφή και ούτω καθεξή. Και εδώ έχω την εντύπωση ότι δεν είμαστε στο ύψος των περιστάσεων όσον αφορά τα δικαιώματα, την προστασία και εγγυήσει που πρέπει να προσφέρουμε στους συμπολίτε μας. Έχουμε μάλιστα πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Και ως ε, δημοκρατικό όργανο θα πρέπει να ενεργήσουμε, να δράσουμε, γιατί είμαστε ένα αντίβαρο στην εξουσία. Είμαστε ένας θεσμός που πρέπει να ξεπεράσει όλες τις κριτικές ώστε να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των εργαζομένων, των ανθρώπων και των καταναλωτών. Και εδώ ε, πιστεύω και φοβούμε πως είναι πολύ αργά, έχουμε πλέον γονατίσει, δεν μπορούμε πια να στηρίξουμε ε, το, παρά μόνο το βιομηχανικό τομέα και αυτό θα γίνει εις βάρος των συμπολιτών μας. Βιαζόμαστε, βιαζόμαστε να εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία, αυτή τη μεγάλη εταιρική σχέση και έχω την εντύπωση πως το Κοινοβούλιο εδώ θα χάσει πολύ περισσότερα από όσα πιστεύει, ε, κυρίως όσον αφορά την, την αξιοπιστία του και την εικόνα του. Θα θεωρηθεί ως ένα αδύναμος θεσμός. Υπάρχουν λοιπόν κάποια σημεία που θέλω εδώ να τονίσω, ειδικά όσον αφορά αυτή την κοινή επιτροπή τη μειχτή μάλλον επιτροπή που ε, έχω την εντύπωση ότι πόρο απέχει από ένα δημοκρατικό σύστημα πρόκειται για μια πέμπτη εξουσία στην ουσία που θα ασχολείται με την νομοθεσία δεν θα είναι μόνο οι, οι υπάλληλοι που θα συμβουλεύουν θα υπάρχει και μια πέμπτη εξουσία αυτή των λόμπι και εδώ δεν είμαι καθόλου σύμφωνη ε, έχουμε στην Ευρώπη το 90% των πολιτών που ε, θίγονται από την ζωή των βιομηχανιών και του εμπορίου. Άρα λοιπόν η ΣΕΤΑ θα είναι κομμάτι της δημοκρατίας μας και της καθημερινής μας ζωής. Αν είναι λοιπόν εις βάρος μας, θα είναι εις βάρος όλων μας. Η διαιτησία δεν νομίζω πως είναι καλή λύση, γιατί για την επιλογή των δικαστών εκεί. Επανειλημμένως προσπαθήσαμε να στραφούμε προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να το επιβεβαιώσουμε κατά πόσο αυτό το σύστημα συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ε, ειλικρινά εγώ δεν έχω ιδέα πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα, αν θα είναι βιώσιμο, αν θα σταθεί στο ύψος των 500 διαβουλεύσεων που είχαμε ε, ας πούμε στη διάρκεια των μεγάλων δημόσιων ε, διαβουλεύσεων και συζητήσεων. Έχουμε την εντύπωση λοιπόν πως οι αμερικανικές εταιρείες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτό για να περάσουν μέσω του Καναδά στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να εξηγηθούν διάφορα πράγματα, διάφορες επεξηγήσεις γιατί διαφορετικά θα χαθούμε σε έναν πολιτικό και νομικό ε, λαβύρινθο. Ξέρω πως αυτή η συμφωνία θα χρησιμεύσει ως πρότυπο για τη μελλοντική συμφωνία με τη Σιγκαπούρη και πρέπει να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε το σύστημα. Αυτό έχουμε στείλει σχετικές τροπολογίες. Ε, για τους πρασίνους. Ε, τώρα έχουμε την Χάιδη Χάουταλα. Καλώς ορίσατε εδώ, σε αυτή την επιτροπή μας. Ε, και τώρα σας δίνω και αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ. Επίτροπε, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτές οι συνολικές περιεκτικές συμφωνίες διεθνούς εμπορίου, οι οποίοι ξεπερνούν τα ζητήματα των δασμών, είναι το μέλλον. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την ισπανική διερμηνία. μιλάει ο, ο αλλά υπάρχει κάποιο πρόβλημα θορύβου στην, στην Ισπανία ε, βουλευτή. Ίσως υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα με την καμπίνα. Okay, um, Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, έλεγα ότι δεν αμφιβάλλω ότι το μέλλον βρίσκεται σε αυτές τις ε, συμφωνίες που είναι πλήρεις, περιεκτικές ε, και συμπεριλαμβάνουν πολλέ πτυχέ του διεθνούς εμπορίου με μεγαλύτερη εναρμόνιση της νομοθεσίας. Αλλά Α αναγνωρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε νερά χαρτογράφητα και άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς κινούμαστε. Όταν ξεκινούμε να συνάπτουμε τέτοιου τύπου συμφωνίες όπως αυτή που τίθεται ενώπιόν μας. Και με αυτήν τη λογική εγώ υπέβαλα μια τροπολογία, την έκτη, με την οποία ζητάτε η αναστολή της ε, επικύρωσης της συμφωνίας για πέντε ε, μήνες. Γιατί εγώ πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ακολουθήσει τη δικιά τις δικές του αρμοδιότητε και προτεραιότητες, να ασκήσει αυτές τις αρμοδιότητες, ιδίω όσον αφορά την ε, ε, Κοινή Επιτροπή. Ε, χαίρομαι που ο συνάδελφος Μόιζα έθεσε αυτά τα ερωτήματα σε εσά και χαίρομαι επίσης που και εσείς κύριε Επίτροπε απαντήσατε. Όμως, η απάντηση που λάβαμε ενθαρρύνει την άποψή μου, ενισχύει την άποψή μου, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ανησυχεί από τι αρμοδιότητε που δίνονται σε αυτή τη μεικτή επιτροπή να τροποποιεί παραρτήματα. Είπατε ότι κάποια από αυτά τα παραρτήματα δεν είναι ε, ευαίσθητα, δεν είναι κρίσιμα. Όμω αυτό είναι ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί, θα δούμε. Ε, και αυτή η Εμικτή Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί. Είπατε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την πλήρη εξουσία με βάση τη Συμφωνία της, ε, για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέτει τους κανόνες όσον αφορά την προστασία, την εμπορική προστασία. Όμως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έχει καμία κανένα ρόλο να υποπτεύει, να ελέγχει τι όποιε αλλαγέ θα αποφασίζει και θα υλοποιεί αυτή η κοινή επιτροπή. Ε, γνωρίζετε ότι οι συζητήσει ε, για τη διαθεσμική συμφωνία ε, έχουν διαρκέσει επί μακρόν και κυρίω ένα σημείο στο οποίο υπάρχει διαφωνία είναι η παράγραφο 40 αυτή τη διαθεσμική συμφωνία, που αναφέρεται στο δικαίωμα πληροφόρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο, του Ευρωπαϊκού, να συστημίσω, θεωρεί ότι αυτή η μεικτή επιτροπή έχει τόσο μεγάλη εξουσία, τόσο μεγάλη σημασία, που ζήτησε και πέτυχε να χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο για να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σε αυτή τη μεικτή επιτροπή. Η δήλωση 99 που του Συμβουλίου ε, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς όμως από την πλευρά μας δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι πρέπει να φτάσουμε στην ολοκλήρωση και την υλοποίηση τη διαθεσμική συμφωνία, έτσι ώστε να μπορεί να ασκήσει τον εποπτικό του ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την Επίτροπο που ήρθε σήμερα εδώ. Η θέση μας ως ομάδα είναι σαφής. Έχουμε, την έχουμε πει επαναλημμένως και εξασφάλιση για μας θα πρέπει να είναι ε, πιο σίγουρη, γιατί Φαίνεται να είναι η ΣΕΤΑ συνθήκη, αλλά στην ουσία είναι μια θεσμική μεταρρύθμιση. Αυτό το θέλουν οι πολυεθνικές και οι μεγάλοι επενδυτές. Επιπλέον περιλαμβάνει τις ίδιες αμφισβητήσιμες ρήτρες Ε, που προτάσουν τις δυνατότητες ε, των πολυεθνικών, των ομίλων να ε, προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα και δεν θα είναι μόνο οι καναδικές πολυεθνικές αλλά και το 80% των αμερικανικών πολυεθνικών που έχουν ήδη θυγατρικές στον Καναδά. Δυστυχώ, όπως και σε προηγούμενη περίπτωση της TTIP, οι εταιρείε οι οποίες θα στραφούν κατά των κρατών θα, θα το κάνουν, ή τα κράτη θα αντισταθούν μάλλον με τα χρήματα των φορολογούμενων, που θα είναι όλο και φτωχότεροι. Προετοιμάζεται λοιπόν ε, η αγορά μας να πλημμυρίσει με κρέας με ορμόνες, με διάφορα προϊόντα. Λέει και σήμερα μας είπατε πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από τη ΣΕΤΑ. Μόνο το 1% όμως αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν εμπόριο πυρατλαντικό και ε, τέτοιου είδους γραφειοκρατική διαδικασία δεν θα βοηθήσει να επεκταθούν περισσότερο. Το είδος ε, της, ε, δε, της διανομής που υπάρχει είναι τελείως διαφορετικό. Δεν θα βοηθήσει η ΣΕΤΑ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μόνο τις μεγάλες άλλες σίγουρα θα εξυπηρετήσει. Εξάλλου η ΣΕΤΑ θα αρχίσει να ισχύει χωρίς να περάσει από την έγκριση των Εθνικών Κοινοβουλίων θα ε, αρκέσει να το υπερψηφίσει εδώ το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό. Πιστεύω πως οι πρόσφατες διαβουλεύσεις ε, δείχνουν ότι ε, ο κόσμος θέλει τη διαχείριση της παγκοσμιοποίησης και όχι την νομική της δίθεν ρύθμιση. Δυστυχώς ακολουθήθηκε λάθος διαδικασία. Η ΣΕΤΑ βέβαια κάπως ε, καλοπίστηκε, αλλά παρόλα αυτά στην ουσία συνεχίζει να αποτελεί μια επίθεση κατά των βασικότερων δικαιωμάτων. Εμείς θα αντισταθούμε και θα στηρίξουμε αυτό που μας έχουν ζητήσει οι πολίτες. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρία Μαρία Αρένα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για το γεγονό ότι ενθαρρύνατε ε, τον διάλογο που είχαμε μέχρι στιγμή για την ΣΕΤΑ και επίση να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πάντοτε παρευρίσκεστε δεν δίνετε απαντήσει στα ερωτήματά μα. Είναι σαφέ ότι δεν είναι εύκολο αυτό το έργο είχατε να διαπραγματευτείτε μια συμφωνία η οποία συμφωνήθηκε αρχικά με την Επιτροπή Μπαρόσο και τον Επίτροπο Εμπορίου, την τότε Επίτροπο Εμπορίου, την κυρία Ντικούχτ, και την προηγούμενη κυβέρνηση του Καναδά, τον κύριο Χάρπερ. Ε, καταφέραμε να επιτύχουμε επιτυχίες, να επιτύχετε βήματα, όπως για παράδειγμα ε, το ISDS που αντικαταστάθηκε με το δικαστήριο. Όμως είμαστε ακόμα στα μισά του δρόμου. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί μας ε, λέτε ότι θα πρέπει να υπερψηφίσουμε μία συμφωνία η οποία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ε, όταν έχουμε ήδη μία χώρα η οποία έχει αποφασίσει να μην την κυρώσει, ως έχει, μιλώ προφανώς για το Βέλγιο. Μας ζητάτε λοιπόν να αποδεχτούμε ένα κείμενο νομικό το οποίο δεν θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή γιατί υπάρχει ήδη μία χώρα η οποία έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να το κυρώσει. Άρα δεν θα ήταν πιο λογικό να, ε, ε, περιμένουμε κι άλλο. Τίθεται επίση το ζήτημα τη συμβατότητα αυτού του νομικού κειμένου με το ε, ευρωπαϊκό νομικό κεκτημένο. Ε, στον υπόθεση με τη Σιγκαπούρη, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διευκρίνησε ότι πρόκειται για μεικτή συμφωνία, συμφωνία μεικτή αρμοδιότητα, επομένω δεν έδωσε. Ε, δεν, δε, συμφώνησε με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ζητήσουμε τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Νομοδότησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το κατά πόσον το σύστημα ISDS, το σύστημα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είναι συμβατό με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη. Είπατε επίσης ότι η προστασία του περιβάλλοντος και των ε, ε, εργατικών δικαιωμάτων θα είναι νομικά δεσμευτική. Όμως αυτό δεν ισχύει σήμερα. Είναι κάτι το οποίο το ζητούν οι πολίτες μας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης η COP21 υπεγράφει συμμετέχουμε στη διαδικασία της COP22 και τίποτα δεν διασφαλίζει την τήρησή τους και, τη και την, και την ε, προστασία τους με βάση τη ΣΥΤΑ ή αυτήν την συμφωνία. Επομένως δεν είναι μια συμφωνία του 21ου αιώνα όπως μας λέτε. Είδατε ότι είχαμε διαμαρτυρίες των αγροτών σήμερα μπροστά από την κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί? Γιατί ακριβώς δεν δέχονται αυτή την απορρίθμιση της αγοράς. Όλες αυτές οι συμφωνίες όπως η ΣΥΤΑ και άλλες οδηγούν σε ακόμη μεγαλύτερη απορρίθμιση της αγοράς. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτό δεν το επιθυμούν καθόλου οι πολίτες μας. Η κυρία Σαϊφή, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε σήμερα εδώ, την παραμονή αυτής της σημαντικής ψηφοφορίας και σας ευχαριστώ που ήσασταν διαθέσιμοι για μας και για να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω άλλη μια φορά ότι για μας η ΣΕΤΑ είναι μια ενδιαφέρουσα συμφωνία που προσφέρει ευκαιρίες. Εμείς έχουμε επανειλημμένα ρωτήσει την Επιτροπή και έχουμε πετύχει δεσμεύσεις για διάφορα σημεία. Εμείς θέλουμε ελεύθερη συναλλαγές που θα απαντούν στην αμοιβαιότητα και στο αμοιβαίο όφελος. Όσον αφορά τις ελεύθερες συναλλαγές και τις εμπορικές συμφωνίες, δεν θα κυρώσουμε συμφωνίες ε, πάση θυσία με οποιοδήποτε τύπημα, τίμημα και είπαμε ότι αυτές οι συμφωνίες δεν θα πρέπει να πλήξουν τις αξίες μας ούτε τις επιλογές μας τις κοινωνικές ή το δημόσιο τομέα, τη γεωργία. Θα ήθελα ωστόσο να εκφράσω την ανησυχία μου, διότι γύρω από τη συζήτηση για την ΣΕΤΑ ε, και τα όσα έγιναν με τη TTIP, ε, βλέπουμε πολύ καλά στη κοινή γνώμη υπάρχει μια γενικότερη αμφισβήτηση όσον αφορά το διεθνές εμπόριο. Έχει γίνει πραγματική συζήτηση πλέον αυτό το Σαββατοκύριακο και πιστεύω πως όλοι οι βουλευτές το γνωρίζουν. Είχαμε διάφορες ε, και πολλές και διάφορες διαδηλώσεις και στις όλες μας τις πόλεις και μάλιστα στις πόλεις μας ε, είχαμε, ε, είχαν μπροστά τους ε, τις φωτογραφίες μας με το όνομά μας και έδειχναν τους ευρωβουλευτές που ετοιμάζονται να υπερψηφίσουν τη ΣΕΤΑ. Πολύ ανησυχητική φάση έχουμε περάσει. Πώς λοιπόν σήμερα εμείς ε, τι θα κάνουμε για να μπορέσουμε να μάθουμε στον κόσμο, να τον πείσουμε και να γίνει μια γενική συζήτηση για το διεθνές εμπόριο. Να εξηγήσουμε όπως το κάνουμε ήδη πώς ε, ανάπτυξη θα πρέπει να την αναζητήσουμε εκτός Ευρώπης, ε, ότι δεν μπορούμε να κλεινόμαστε στον εαυτό μας, ειδικά τη φάση που ο κύριος Τραμπ ε, κάνει τις δηλώσεις του δεξιά και αριστερά. Θα κλείσουμε λοιπόν τα σύνορα, θα κάνουμε προστατευτισμό. Εγώ θέτω την ερώτηση και πιστεύω πως ε, ίσως θα πρέπει μετά από την ψήφο για αυτή την ε, συμφωνία να μπορέσουμε να ε, δείξουμε στον κόσμο, να τον μάθουμε τι ακριβώς συνέβη, να τον ενημερώσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σούστερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τη συμφωνία, όμως προσπαθήσαμε πολύ τα τελευταία δύο χρόνια για να φτάσουμε στο ε, τέλος αυτού του στόχου. Σίγουρα αυτά τα δύο χρόνια δεν έφτασαν και ε, να πω όμως ότι στο θέμα των επενδύσεων έχουν γίνει πάρα πολλά, έχουν αποσαφενιστεί πολλές ασάφειες. Μετά, πολύ μεγάλη σημασία έχει ο ε, κώδικας δεοντολογίας των δικαστών. Δεν είναι ακόμα έτοιμος. Παρομοίως και για ε, τις ε, κυρώσεις εις βάρος των εργοδοτών εάν δεν σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ε, δεν υπάρχει μεγάλη σαφήνεια επίσης το τι θα γίνει με την επίλυση διαφορών, ιδιαίτερα στην περίπτωση των επανακρατικοποιήσεων επιχειρήσεων. Ε, τώρα, να πω πως ε, φυσικά και έχω εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως ε, ως Ευρωβουλευτής πρωτού κύρωσω κάτι θα πρέπει να γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες και στην προκειμένη περίπτωση θα ήθελα να γνωρίζω το τι συμβαίνει με αυτόν τον κώδικα διοντολογίας, αν έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Η συμφωνία ΣΕΤΑ σίγουρα δεν θα έχει τρομερές επιπτώσεις τόση στην παγκοσμιοποίηση δεν θα την βοηθήσει, δεν θα την αποτρέψει. Όμως η απελευθέρωση των αγορών είναι μια λογική την οποία ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια. Αυτή η λογική όμως έχει οδηγήσει και σε προβλήματα περιβαλλοντικά αλλά και σε συζήτηση για το πώς μπορούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, για το ε, τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά με τις ανισότητες, ε, τις κοινωνικές, τις εργασιακές που έχουν παρα, ε, τηρηθεί. Και σίγουρα αυτή η απελευθέρωση είναι το πρώτο μέλημά μας όταν συζητάμε αυτή τη συμφωνία. Τώρα, Πιστεύω πως ε, σίγουρα δεν είναι ε, παρκή η συμφωνία αυτή, διότι δεδομένων των ε, πρόσφατων εξελίξεων πολύ φοβάμαι πως τα πράγματα θα επιδεινωθούν. Αυτός ο προστατευτισμός θα διεγκωθεί και θα οδηγήσει σε περαιτέρω κρίσεις. Μάλιστα σε κρίση που πολύ φοβάμαι θα μοιάζει με αυτή της δεκαετίας του 30. Ανεξάρτητα τώρα με το τι θα γίνει ε, με τη συμφωνία ΣΕΤ, αν θα ψηφιστεί ή όχι, πιστεύω πως βρισκόμαστε ενώπιον μιας άλλης ε, ε, διάστασης, μιας αλλαγής και θα πρέπει να ξανασκεφτούμε το πώς θα συμπεριφερόμαστε απέναντι στους δύο μεγαλύτερους εταίρους μας, τις Ηνωμένε Πολιτείε δηλαδή και την Κίνα. Αυτές είναι ερωτήσεις οι οποίες πρέπει να απαντηθούν άμεσα και να συζητηθούν εντατικά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φιέλνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αναρωτιέμαι αν θα έπρεπε να δώσουμε ένα βραβείο σήμερα. Ένα βραβείο, το βραβείο ΣΕΤΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να δώσουμε ένα μπουκάλι σαμπάνια. Εγώ προσωπικά θα βραβεύσω με ένα μπουκάλι σαμπάνια σε όποιον δώσει μια νέα πρόταση, μια, ένα νέο επιχείρημα υπέρ τη σύναψη αυτή τη συμφωνία. Είναι η έκτη φορά που γίνεται αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Στις 12 ε, Οκτωβρίου είχαμε πάλι μια ανταλλαγή απόψεων με ενδιαφερόμενους, ε, Νοεμβρίου, πάλι άλλη μία, Δεκέμβριο στο Στραμβούργο, ανταλλαγή απόψεων με την νομική υπηρεσία, 9 ε, Δεκεμβρίου πάλι ανταλλαγή απόψεων, σήμερα πάλι το ίδιο, έχουν γίνει πολλές ε, μεικτές συνεδριάσεις. Πήγαμε δύο φορές στον Καναδά Στείλαμε προσωπία. γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι όποιο από εσά βρει ένα καινούργιο επιχείρημα υπέρ τη συναψυμφωνία αξίζει βραβείο. Όμω πιστεύω πω ε, πρέπει να συζητήσουμε κι άλλο. Δεν μα φτάνει ε, αυτό η προσπάθεια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα ήθελα να υπάρξει μια ε, αναβολή. Τα επιχειρήματά μου δεν είναι τα ίδια με εκείνα της ε, κυρίας Επιτρόπου διότι σίγουρα πιστεύω πως αυτή η συμφωνία είναι καλή, πάρα πολύ καλή. Εάν πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτή η συμφωνία θα δώσει καλύτερη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον Καναδά από εκείνη την πρόσβαση που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τότε μπράβο. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή αναφέρεται στη συμφωνία ναύτα λέγοντας ότι τέλος πάει, θα την πετάξει στα σκουπίδια. Γι' αυτό λοιπόν είναι επίσης είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή να συναυτεί αυτή η συμφωνία. Αν δεν μπορούμε να την ολοκληρώσουμε, ποια συμφωνία θα είναι αυτή που μπορούμε να κάνουμε. Όμως, με όλες αυτές τις συζητήσεις που έχουν γίνει, νομίζω πως όλοι οι ε, εταίροι μας στον κόσμο αναρωτιούνται εάν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε business μαζί τους, αν θέλουμε να συνεργαστούμε. Και στη Βραζιλία αυτό ε, μάλλον θα λένε. Δεν νομίζω πως πρέπει να μας απασχολεί το τι θα κάνει ο Τραμπ στις ΗΠΑ προς το παρόν, ή τουλάχιστον τον καθημερινό κοινό άνθρωπο δεν τον απασχολεί. Αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει όμως είναι το πώς εμείς θα δεσμευτούμε για να κάνουμε τη διαφορά στο εμπόριο. Και το πώς θα το κάνουμε αυτό θα ε, το κάνουμε ε, ολοκληρώνοντας και συνάπτοντας τη συμφωνία αυτή. Και ποια είναι αυτή, το αυτοβραβείο που είπατε, ένα μπουκάλι σαμπάνιας. Θέλετε να σας πω και τη μάρκα της σαμπάνιας. Ε, εντάξει, ευρωπαϊκή θα είναι. Δικιά μας. Θα είναι και pop. Πολύ ωραία. Τέλεια, τέλεια. Κύριε Κράσφελτερ, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Μάλιμστρομ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, που είστε διαθέσιμοι στην Επιτροπή μας για να απαντήσετε τις ε, ερωτήσεις μας. Βρισκόμαστε ενώπιν μιας νέας εποχής πράγματι με τη σύναψη αυτής της συμφωνίας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε τι ακριβώ έχει γίνει μέχρι τώρα. Να κάνουμε έναν απολογισμό, να δούμε πού μα έχουν οδηγήσει οι διαπραγματεύσει. Είμαστε πιστεύω στο σωστό δρόμο, όμω θεωρώ πω δεν έχουμε φτάσει τόσο μακριά όσο θα έπρεπε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο στάδιο που θα μπορούσαμε να πούμε τέλο η συμφωνία ολοκληρώνεται. Έχουν αποδειχθεί τα προβλήματα που συναντήσαμε και οι διευκρινήσει που δώσατε, για παράδειγμα για αυτή τη μεικτή επιτροπή ΣΥΤΑ, είναι σίγουρα πάρα πολύ χρήσιμες. Όμως ε, διαρωτώ με εάν δεν θα ήταν καλύτερο όλες αυτές οι διευκρινήσεις να πάρουν τη μορφή ενός δεσμευτικού πρωτοκόλλου το οποίο θα ε, δημοσιοποιηθεί. Τονίζω το νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα. Μετά, ε, α, αυτές τις επιφυλάξεις δεν τις έχουμε μόνο για την ε, μυστική συνεργασία, αλλά και ο Ιωάχημ αναφέρθηκε στο επενδυτικό ε, θέμα, στην επίλυση διαφορών, στο, σε, στο κεφάλαιο που θα αφορά τη βιωσιμότητα. Εδώ νομίζω πως ε, υπάρχουν πολλές βελτιώσεις τις οποίες δεν έχουμε καταφέρει να φέρουμε στο κείμενο, οι οποίες όμως είναι αναγκαίες. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν αυτά τα προβληματικά σημεία παραμείνουν όσα έχουν προβληματικά και δεν επιληθούν, τι θα γίνει. Θα μπορέσουν τα κρατημέλη να κυρώσουν τη συμφωνία αυτή. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνω τώρα τον κατάλογο των ομιλητών. Άλλοι 7 περιμένουν να μιλήσουν. Ο κύριος Όμπερμαϊερ στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και να σας συγχαρώ επίσης και για την επανεκλογή σας. Νομίζω πως ε, δεν χρειάζεται βιασύνη στις συζητήσεις μας για τη Συμφωνία ΣΕΤΑ. Σίγουρα έχουν γίνει πολλές ε, προτάσεις που βελτιώνουν το κείμενο, που βελτιώνουν το αρχικό κείμενο, που πιστεύω πως έχει οριμάσει αρκετά αυτό το κείμενο. Από την άλλη όμως η πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή η εκλογή του Τραμπ δηλαδή και πολλά άλλα μας οδηγούν σε σκέψεις για το τι θα γίνει στο μέλλον. Είπε ο Τραμπ ότι θα καταργήσει τη Συμφωνία Ναύτα. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε να εκτιμήσουμε, να αποτιμήσουμε την κατάσταση και να δούμε ε, ποιες θα είναι οι συνέπειες μιας ενδεχόμενης ακύρωσης της συμφωνίας ναύτα. Τι θα γίνει με τις θηγατρικές αμερικανικές εταιρείες στον Καναδά, πώς αυτό θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή αγορά αλλά υπάρχουν και κάποια πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που έχω τουλάχιστον εγώ. Ε, στα πλαίσια της αριθμιστικής συνεργασίας δεν βλέπουμε κάποια ε, βελτίωση, δεν βλέπουμε κάποια σαφή ρύθμιση, σαφή βελτίωση της εφισταμένης κατάστασης. Βλέπω πως υπάρχει κίνδυνος να αποδυναμωθεί η νομοθετική μας εξουσία εδώ. Μετά, σε ό,τι αφορά το δικαστήριο, το πενευτικό δικαστήριο. Εδώ πιστεύω πως ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε μια τέτοια περίπτωση διαφωνίας και πως ε, δεν θα λαμβάνονται υπόψη παραβιάσεις που θα γίνονται από μεγαλύτερους ομίλους. Μετά, να μην ξεχνάμε και την πίεση που ε, ασκείται για να ολοκληρωθούν γρήγορα οι διαπραγματεύσεις και να συναυθεί η συμφωνία. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, γίνεται δημοψήφισμα για τη συμφωνία ΣΕΚΑ έχουμε αφήσει στους πολίτες την τελευταία λέξη και πιστεύω πως αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σίλβα Περέιρα έχει το λόγο. Εγώ πιστεύω πως αυτό η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά είναι στρατηγική σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή την εποχή που από ό,τι φαίνεται είναι εποχή προστατευτισμού, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται και για νέες μορφές ανταγωνισμού για το, που αφορούν το μέλλον των παγκόσμιων εμπορικών ροών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να δώσει οικονομική απάντηση που να είναι στο ύψος αυτών των προκλήσεων, ούτε απομόνωση, ούτε η αναβολή είναι απαντήσεις. Η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε θέση να πει ότι ήταν πολύ απαιτητικό με τους διαπραγματευτές για ε, για να μπορέσει να ε, προστατεύσει τους πολίτες. Όμως, ε, επίσης, έχει την ευθύνη, εφόσον οι διαπραγματευτές φέραν καλό αποτέλεσμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και η Ευρωπαϊκή η Διαπραγματευτική Ομάδα της οποίας ηγήθηκε ο Μάουρο Πέτρος και το, όσο και η νέα κυβέρνηση του ε, Καναδά έφτασαν σε μια συμφωνία που, δεν είναι απλά ισορροπημένη από πολλές απόψεις είναι μια προοδευτική συμφωνία που προσδιορίζει ένα καλό πλαίσιο, ένα καλό σχήμα για το μέλλον του διεθνούς εμπορίου. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν την αλήθεια και πιστεύω πως η συμφωνία αυτή αξίζει την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και άρα και τη θετική ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Thanks a lot. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Σάντζεσ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, που είστε σήμερα εδώ. Εγώ αυτή τη σέτα τη βλέπω, μου θυμίζει το ρούχα του αυτοκράτορα, αυτό το παραμύθι. Ε, είναι μια εμπορική συμφωνία που είναι εντυμένη με τα ρούχα της απασχόλησης, της ευημερία, της αύξησης ε, των στάνταρ των εργασιακών, των περιβαλλοντικών. Είμαι όμως αυτό το ρούχο που φοράει εδώ μέσα, γιατί έξω δεν το βλέπει κανένας αυτό το ρούχο. Δεν το βλέπουν ούτε τα συνδικάτα, ούτε οι ενώσεις, ε, ούτε οι προμεσαίες επιχειρήσεις, ούτε η ΜΚΟ, ούτε η κοινωνία των πολιτών, ούτε οι γεωργοί. Δεν το βλέπουν πάνω από 3.000 δήμοι σε ολόκληρη την Ευρώπη, ούτε καν η Επιτροπή Απασχόλησης σε αυτό το, το, το, το κοινοβουλίο δεν το βλέπει το ρούχο αυτό έχουν αρχίσει και χτυπάνε όλα τα καμπανάκια, ειδικά στην Επιτροπή Απασχόλησης, ενώ εδώ φαίνεται να, να, μην ακούμε τίποτα. Θα πρέπει ωστόσο να τους ακούμε καλύτερα. Και εμείς έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά στο τι λέει ο κόσμος στο, και θέλω να οι σοσιαλιστές που, που ανακοίνωναν αυτή τη ρήξη της μεγάλης συμμαχία πριν από τις εκλογές του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου είναι η ώρα να το αποδείξουν ότι υπάρχει όντω ρήξη. Ε, ακούμε τι γίνεται λοιπόν ε, στο δρόμο, στους δρόμους, οι διαδηλώσεις. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν μια, ένα σοβαρό πολιτικό σφάλμα γιατί αυτό που βλάπτεται περισσότερο είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα. Η εικόνα που έχει ο κόσμος για μας. Είμαστε σε μια κατάσταση εξαιρετικά κρίσιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όσον αφορά την εικόνα μας προς τον κόσμο. Αν μας βλέπει κοντά του, αν θεωρεί ότι είμαστε απόμακροι και απομακρυσμένοι και ο κόσμος τελικά, αυτοί που ψηφίζουν και αυτοί που δεν θα ψηφίσουν ακόμα είναι τα αφεντικά μας. Θα έπρεπε εμεί να ανοίξουμε λίγο περισσότερο τα παράθυρα και τις πόρτες αυτών των κτηρίων, να ανανεώσουμε λίγο τον αέρα και να αφήσουμε αυτοί που υποφέρουν και ζουν τις πολιτικές που εμείς ε, ψηφίζουμε να μας πούν ακριβώς ε, τι ζουν καθημερινά. Εμείς δεν θέλουμε να αφαιρέσουμε ε, εξουσίες από τα κυρίαρχα κοινοβούλια. Θα είναι όμως αυτή μια συνέπεια αυτή τη ΣΕΔΑ και αν συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό και να το υπερψηφίσουμε θα δώσουμε λαβή ακόμη περισσότερο σε αυτούς που θέλουν να διαλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πιστεύουμε την Ευρώπη και είμαστε βαθιά ευρωπαϊστές, είμαστε ευρωπαϊστές όμως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Εγώ αύριο θα καταψηφίσω. Δεν είμαι κατά του διεθνούς εμπορίου, ούτε κατά το διεθνούς σχέσεων ωστόσο. Είμαι κατά αυτού του μοντέλου που βλάπτει τους ανθρώπους, βλέπει τα άτομα και προτάσει τα κέρδη λίγων, ολίγων Ευρωπαίων και γι' αυτό και κανείς από αυτούς δεν λέει ότι ακολουθούμε τον κακό δρόμο, τον λάθος δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ροντρίγκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. una vez, no van a dar el εγώ θέλω να πω τα εξή. Τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί. Η ΣΕΤΑ είναι μια καλή συμφωνία, αλλά στην ακατάλληλη στιγμή. Ακατάλληλη στιγμή είναι πολλές φορές αυτοί που είναι κατά της παγκοσμιοποίησης, ε, που είναι συνέπειες των εθνικών μας πολιτικών που δεν καταπολεμούν την ανισότητα, τη λάθος κατανομή πλούτου και δεν δημιουργούν μια βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα αυτά τα ρίχνουν στις εμπορικές συμφωνίες και, αν έχει κάνει... και λένε ότι με αυτό καταψηφίζουν την παγκοσμιοποίηση και άρα και το διεθνές εμπόριο. Αν βελτιωθούν ε, οι οικονομικές συνθήκες υπό τις οποίες παράγονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες υπό αυτή τη συμφωνία, ναι, εντάξει, την εγκρίνουμε. Υπάρχουν, μια, υπά, υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, τις καταλαβαίνω, μια εμπορική συμφωνία ποτέ δεν θα είναι τέλεια, πάντοτε θα έχουμε κάποια στοιχεία που θα μπορούμε να βελτιώσουμε και κάποιες λογικές αμφιβολίες. Το σημαντικό όμως είναι και πού μας πάνε τα βήματα που ακολουθούμε. Και σε αυτή τη συγκυρία εγώ διερωτώ. είναι καλύτερο να υπάρχει σύστημα διατησίας ή ένα επενδυτικό δικαστήριο που θα παίρνει όσον αφορά το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κανείς δεν το επικρίνει γιατί αυτό είναι το πρότυπο που ακολουθεί. Είναι καλύτερο ο Καναδάς τώρα που έχει ήδη υπογράψει 7 συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας ή όχι. Είναι καλύτερο να δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεργαστούμε για να γίνουν οι πολυμερές στο δικαστήριο το επενδυτικό ή όχι. Ε, ε, εγώ πιστεύω πως ναι. Πιστεύω ότι αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή, που είναι εξαιρετικά δύσκολη φάση, με την ε, πρόοδο της του προστατευτισμού και της δημαγωγίας, εγώ υπερασπίζομαι περισσότερο από ποτέ την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αρχές της και τις αξίες της, που ναι πάντα θέλει να προχωρήσει με τις πρακτικές της και ότι αυτό το, και πιστεύω πως αυτή η συμφωνία είναι ένα βήμα μπροστά και θα πρέπει να χρησιμεύσει όσον αφορά σε ένα κεφάλαιο βιώσιμης ανάπτυξης που θα έχει αναγκαστικά και οπωσδήποτε περιλάβει την, τον υποχρεωτικό της χαρακτήρα. Και θέλω να κάνω και μια ερώτηση. Τι μάθαμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή, αυτή την πορεία. Υπάρχουν πολλές πτυχές μιας συμφωνίας, ε, πολύ γενικές, που θα πρέπει να γίνουν πραγματικά προσπάθειες για να ανταποκριθούμε και να καλύψουμε τις διάφορες αμφιβολίες και ανησυχίες. Θα πρέπει από αυτό να μάθουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια συμφωνία προοδευτική όπως είναι τούτη εδώ. Ευχαριστώ. Άρτσο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύρια Μάλμστρομ. Θα συμφωνήσω και εγώ με τους προηγούμενους συναδέλφους και θα πω ότι αυτές οι πολύ <laughs> συχνές ανταλλαγές απόψεων ε, ήταν δυνατές χάρη και στη δική σας παρουσία. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε μια εταιρεία, στην ε, ε, Bombardier. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη καναδική εταιρεία η οποία έχει πολλές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κινδυνεύουν να χαθούν λοιπόν αυτές οι θέσεις ε, με τις τελευταίες εξελίξεις. Και αυτή η απώλεια θέσεων εργασία σας θα πλήξει πάρα πολύ τις περιοχές τις οποίες αφορά. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θέλω να ρωτήσω, πώς θα βοηθήσει η συμφωνία ΣΕΤΑ να κρατήσω τη δουλειά μου σε αυτή την περίπτωση. Ποιε είναι οι διατάξεις της συμφωνίας αυτής που αφορούν ζητήματα περιβαλλοντικά, ζητήματα εργασιακά. Πώς μπορούν να κρατήσουν υπόλογους τους ε, υπεύθυνους. Χρειάζεται λοιπόν μια διμερή συμφωνία να είναι και αμφίδρομη, να υπάρχουν συγκεκριμένα ε, κριτήρια, συγκεκριμένα περιβαλλοντικά κριτήρια, συγκεκριμένοι μηχανισμοί προστασίας, τα οποία ε, στοιχεία αυτά θα βοηθούν, θα προστατεύουν τους ε, πολίτες, τους εργαζόμενους όταν συμβαίνει μια τέτοια περίπτωση όπως αυτή της Μπομπαρδιέ. Ε, Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ που αναφερθήκατε και σε αυτές τις πτυχές της συμφωνίας. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε την εντολή του 2009 και να την χρησιμοποιήσουμε, διότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Υπάρχει μεγαλύτερη απελευθέρωση των αγορών κτλ. Όμως τώρα έχω αρκετές σκέψεις και να πω και κάτι. Ίσως εγώ κερδίσω το βραβείο της ε, καινοτόμου σκέψης. Το σύστημα SES e ακολουθεί την ίδια λογική. Δηλαδή, οι επενδυτές θα έχουν την ε, δυνατότητα να προσφύγουν εναντίον των ε, επιχειρήσεων, εναντίον κατών Είναι λοιπόν αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν ο νομοθέτης ή αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει πραγματικά να αλλάξει κάτι, μπορεί με να το κάνει, όμως για τον επενδυτή το σημείο αναφορά σε μια τέτοια περίπτωση ε, διαιτησίας θα είναι η συμφωνία, θα είναι το άρθρο 831. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι το συγκεκριμένο άρθρο 831 πρέπει να το επανεξετάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, και ο κύριος Προύστ και σα ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που για άλλη μια φορά ήρθατε εδώ για να συζητήσουμε για αυτά τα ζητήματα. Σε καμία περίπτωση κανείς δεν μπορεί να σας προσάψει ε, έλλειψη συμμετοχή στον πολιτικό διάλογο. Πάντα έρχεστε και απαντάτε ε, στις ε, αντιρρήσεις μας, στις απορίες μας. Παρά το γεγονό ότι έχουμε συμφημιώσει πρόοδο και έχουμε κάποιες βελτιώσεις. Πιστεύω ότι τελικά αυτοί που επιθυμούσαν να ψηφίσουν κατά θα καταψηφίσουν, γιατί όταν ακούω λεξιλόγιο του τύπου ε, ότι η παγκοσμιοχή είναι διαβολική κτλ. Παρόλο που σέβομαι τις απόψεις κάθε συναδέλφου, πιστεύω ότι με τέτοιου τύπου ε, διατυπώσεις ε, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Έχουμε μια κατάσταση όπου σήμερα ορισμένοι μας λένε ότι αν δεν, δεν επικυρώσουμε τη ΣΕΤΑ η ε, ε, κατάστασή μας θα βελτιωθεί. Δεν ισχύει αυτό. Όμως, εάν έχουμε μία συμφωνία με, όπως η ΣΕΤΑ, μία ε, επιχείρηση όπως η ε, Bombardier η οποία συνεργάστηκε με την Κάλστρομ για να ε, προτείνει να συμμετάσχει σε δημόσιες προμήθειες δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει ενώ αυτή τη στιγμή εάν είχαμε τη ΣΕΤΑ θα μπορούσε να το κάνει. Ούτε η σημερινή κατάσταση μας ε, διασφαλίζει τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης. Ε, όταν βλέπω προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν στη γαλλική αγορά που είναι απλώς μαϊμού και αντιγραφές ε. POP. Επομένως, η ΣΕΤΑ και παρόμοιες συμφωνίες θα μας επιτρέψουν να αντιστρέψουμε την κατάσταση, θα μας επιστρέψουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες να εισχωρήσουν στην καναδική αγορά, κάτι που θα δημιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, θα μας επιτρέψουν να ανοίξουμε ε, την αγορά αυτή. Και επίσης ο όποιο προστατευτισμό επιλέξουμε να ελοποιήσουμε θα είναι ευφυή, θα γίνει με έναν τρόπο στρατηγικό και όχι με τον ανόητο και γενικό τρόπο που επιθυμεί να προωθήσει ο κύριο Τραμπ. Σα ευχαριστούμε. Ο κύριο Φερό. Σα ευχαριστώ. Εγώ διαφωνώ πλήρω με τον Γάλλο συνάδελφο. Εγώ πιστεύω ότι όλα είναι. Όλα θα τα χάσουμε με αυτή τη συμφωνία. Δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε. Ε, έχω την εντύπωση ότι το κλίμα απόψε στη συζήτησή μας είναι πένθυμο. Να σας θυμίσω, είπατε μάλλον ότι όλα τα επιχειρήματα έχουν ακουστεί. Όμως, ας μην ξεχνάμε ότι η συμφωνία αυτή είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που έκανε αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ερχόταν και μας ενημέρωνε μόνο που και που και όταν το επιθυμούσε. 50.000 θέσει εργασία απειλούνται μόνο στη Γαλλία. Εκατοντάδε pop, κυρίω στον τομέα των γαλακτοκομικών του τυριού. Και το σίγουρο είναι, κύριε Πρόεδρε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασθενή και αυτή η συμφωνία δεν θα τη βοηθήσει καθόλου να γιατρευτεί. Έχει ξεκινήσει ένα νέο κύμα αμφισβήτησης από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού πολλών διεθνών συμφοριών εμπορίου. Ο κύριος Τραμπ σήμερα ορθά αντιλαμβάνεται ποια είναι τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα έπρεπε να το χαιρετήσουμε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνίε με την Αυστραλία, με χώρε τη Κεντρική Αφρική, με την Ασία κτλ. κτλ. Κατά την άποψή μου, η ΣΕΤΑ δεν βρίσκεται από τη σωστή πλευρά τη ιστορία και σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του πολιτών καθένα πρέπει να αρθεί στο ύψο των περιστάσεων και κατά την άποψή μου πρέπει να καταψηφίσει αυτή τη συμφωνία. Και τελευταία ομιλήτρια, κυρία Μοσκά. Ευχαριστώ. Εγώ δεν θέλω να προσθέσω τίποτα περισσότερο κατά τη συνθήκης, γιατί πολλοί ήδη τα ανέφεραν και τα έχουμε ήδη συζητήσει στις άριθμες συνεδριάσεις που έχουμε κάνει και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και ξανά. Θέλω μόνο να θυμίσω σε όλους ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο περήφανοι σε σχέση με τη δουλειά που έχει κάνει καθένας από εμά μέσα σε αυτήν την Επιτροπή και αυτή, αυτό το Κοινοβούλιο. Γιατί ποτέ δεν υπήρξε τέτοια συμφωνία που να τροποποιήθηκε τόσο βαθιά χάρη στην εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι ένας ρόλος που ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε να το διεκδικήσουμε διεκδικούμε. Έχουμε ασκήσει μέχρι τέλους τη δικαιώματά μας. Ε, μας μένουν κάποιες διαφορές όσον αφορά την αξιολόγηση σε σχέση με το γεγονός ότι αυτή η εργασία, το κατά πόσο μάλλον αυτή η εργασία ήταν επαρκής ή όχι. Ορισμένοι από εμά επαρκή η οχι ορισμενοι απο εμας θεωρουν οτι ειναι μια δουλεια η οποια θα πρέπει να υπερψηφιστεί, άλλοι όχι, αλλά σίγουρα θα πρέπει αυτό το ρόλο να τον διεκδικήσουμε, γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε κανένα επιχείρημα ενάντια σε αυτούς που λένε πως αυτό το κοινοβούλιο μας δεν έχει καμία λειτουργία. Ταυτόχρονα όμως, ακριβώς όπως οι πολίτες μας λένε, μας ζητούν να λάβουμε υπόψη τις δίκαιες τους και σωστές τους παρατηρήσεις και ανησυχίες, μας ζητούν επίσης να αποφασίσουμε. Γιατί ε, έτσι ώστε στην πολιτική να δοθεί ένας όρος να μην να μην μένουμε χωρίς να λαμβάνουμε απόφαση, γιατί και αυτό δυσαρεστεί τον κόσμο και τον απομακρύνει από τους θεσμούς. Πιστεύω λοιπόν πως πέρα από τις διαφορετικές απόψεις υπάρχουν και μια, κάποιες φάσεις όπου δεν πρέπει πλέον να αναβάλουμε την ψηφοφορία, αλλά να φτάσουμε στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Είναι αλήθεια ότι το συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, 7 χρόνια. Ευκρινήσεις, ε, διαπραγματεύσεις, αναβολές, αλλά νομίζω πως το τελικό αποτέλεσμα είναι πως έχουμε μια πολύ καλή συμφωνία. Έχετε συμβάλει σε αυτή. Τα κράτη-μέλη έχουν συμβάλει και η δημόσια συζήτηση έχει συμβάλει. Και ο κύριος Πετρουτσόνη, που είναι ακόμα εδώ εν ζωή, ζωντανός, <laughs> ε, έχει κάνει τρομερή δουλειά μαζί με την ομάδα του. Και αυτό θέλω να το αναγνωρίσω. Ορισμένοι από εσά θα την κατεψηφίσουν αύριο. Αυτό είναι η δημοκρατία. Αλλά νομίζω πω θα το αναβάλουμε και να το ψηφίσουμε σε 2-5 μήνε δεν θα αλλάξει τη γνώμη σα. Ποτέ δεν θα υπερψηφίσετε αυτή τη συμφωνία. Το να το αναβάλουμε είναι ένα τρόπο να να το αναβάλουμε μόνο. Δεν θα την ξεκαθαρίσει περισσότερο, γιατί νομίζω πως όση και σαφήνεια μπορούσαμε να έχουμε, την έχουμε. Έχουμε πραγματικά ξεπεράσει τους εαυτούς μας. Έχουμε 36 δηλώσεις, έχουμε επιστολές, έχουμε ένα σωρό πράγματα. Και έπειτα θα συμμετέχετε στις λεπτομέρειες για την εκπόνηση των λεπτομεριών του επενδυτικού δικαστηρίου. Πώς θα δουλέψει, το ξέρουμε. Αλλά ε, για τις λεπτομέρειες θα συμμετέχετε. Έπειτα να πω ότι ο κόσμος μας ε, κοιτάει πολύ προσωπικά. Μετά από ότι ε, ο θάψιμο ή την αναβολή της θητή, πολλές χώρες παίρνουν σειρά εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας είμαστε μαζί, ας είμαστε ενωμένοι να δείξουμε πώς κάνουμε καλές συμφωνίες, πώς ε, συμφωνίες που είναι ευκαιρίες για να κερδίσουν όλα τα μέρη. Και δεν θα κερδίσουν μόνο οι λίγοι. Και αν δεν κάνουμε αυτή τη συμφωνία, ε, τότε δεν θα μπορούμε να κάνουμε συμφωνίες. Αυτό θα σημαίνει. Και αυτό θα σημαίνει ότι υποβαθμίζουμε την ε, δημοκρατία. Μιλάμε για τον Καναδά, μια από τις πιο δημοκρατικές ε, χώρες του κόσμου, με σχεδόν καθόλου διαφορά, με πολύ ισχυρό δημόσιο τομέα, με μια προοδευτική κυβέρνηση που μοιράζεται μαζί μας τόσες πολλές από τις αξίες μας. Μα δεν κάνουμε κανένα μια συμφωνία με το διάβολο, δεν υποβαθμίζουμε την ε, δημοκρατία. Κάνουμε μια εμπορική συμφωνία με μια χώρα όπου μάλιστα περιλαμβάνονται τα πάντα από αυτά που ζητήσατε πρώτη φορά. Για εντάξει για το κλίμα, για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για τα εργατικά δικαιώματα δικαιώματα, τα ε, δικαιώματα των ζώων. Όλα όσα έχετε ζητήσει για πρώτη φορά είναι μέσα σε αυτή τη συμφωνία και ανεξάρτητοι ε, ε, ε, εμπειρογνώμονες είπαν ότι είναι η πιο προοδευτική συμφωνία που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Μάλιστα κύριε Κάμπο, γιατί να μην είναι, Κάμπερ, γιατί να μην είναι και μοντέλο για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ελπίζω πω θα είναι λίγο πιο σύντομη διαπραγμάτευση. <laughs> Αλλά θα επανέλθουμε σε αυτή την υπόθεση αργότερα. 40 εκατομμύρια κόσμος είναι ο Καναδάς. Πώ μπορούν να μπορούν να μας απειλήσουν τόσο που να υποβαθμίζουμε, λέει, και να υποσκάπτουμε τη δημοκρατία. 27-28 χώρε, 500 εκατομμύρια κόσμος. Πραγματικά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τίποτα στη ΣΕΤΑ δεν ε, απειλεί τη δημοκρατία. Και θα συμμετέχετε σε όλες τις ε, πιθανές αλλαγέ που μπορούν να προκύψουν και η Μικτή Επιτροπή θα είναι φόρουμ συζήτησης. Εάν υπάρξουν αλλαγέ, θα συμμετέχετε, όπως σας είπα, στις αλλαγέ στην, στην διαπραγμάτευση. Τώρα, για κάποια ευρύτερα ζητήματα. Πώς μπορούμε να, έχουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να τους μιλήσουμε με τους συμπολίτε μας. Όλοι μας πρέπει να συζητήσουμε με τα εθνικά κοινοβούλια, με τις κυβερνήσεις μας, ε, ώστε πολύ γρήγορα να αρχίσουμε να συζητούμε μαζί τους, να τους πούμε ότι υπάρχει άλλος τρόπος να κάνουμε συμφωνίες και όχι μόνο η, κυβέρνηση των ΗΠΑ, του Τραμπ. Δεν ξεκινάμε μια με μια εμπορική συμφωνία. Όπω ξέρετε, πρέπει να έχουμε εντολή από όλα τα κρατημέλη. Σε εκείνη ακριβώ τη στιγμή, όταν ξεκινάμε στη διαπραγμάτευση, τα κράτη-μέλη πρέπει να συμμετέχουν και πρέπει να πηγαίνουν να νικούν τι ανησυχίε, να τι ε, μεταφέρουν στην Επιτροπή, να, ε, να, να, να συζητούν γιατί είναι καλό για τη χώρα μου. Υπάρχουν ευαισθησίε, ναι, ίσω στον τάδε τομέα. Α τα δούμε, α προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτέ τι ανησυχίε. Ναι, υπάρχει, ο κόσμο αλλάζει και πολλοί μένουν χαμένοι σε αυτέ τι αλλαγέ. Ε, Αυτές είναι ο φόβος του, του κόσμου. Και έπειτα για τα εργασιακά ζητήματα. Ναι, λέει και βιομηχανοποίηση, για ρομποτοποίηση, για τεχνολογικέ αλλαγέ, αλλά τα κράτη-μέλη πρέπει να γίνουν καλύτερα στο να αντιμετωπίσουν αυτέ τι αλλαγέ. Να έχουν αναπτυγμένα κοινωνικά συστήματα σε συνεργασία με τι επιχειρήσει, ώστε ο κόσμο να μπορεί να μην φοβάται και να κινείται από μια θέση εργασίας σε άλλη, πράγμα που συμβαίνει σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Άλλε θέσει χάνονται, άλλε δημιουργούνται. Και μια καλή συμφωνία εμπορική μπορεί όντω έτσι να βοηθήσει να χειριστούμε την παγκοσμιοποίηση εφόσον περιέχει κανόνες οι οποίοι είναι προβλέψιμοι. Αυτό πρέπει όντω να το κάνουμε. Δεν υπήρχαν πολλές ερωτήσεις νομίζω, περισσότερα σχόλια άκουσα και εκτιμώ όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε και όλε τι συζητήσει που είχαμε. Ελπίζω πω δεν θα πάψουν να ε, σίγουρα δεν θα πάψουν αν υπερψηφίσετε τη συμφωνία. Θα υπάρξουν και άλλα θέματα σε σχέση με την ΣΕΤΑ πιο συγκεκριμένα και θα συνεχίσουμε αυτή την πολύ καλή συζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Είμαι σίγουρος πως θα παραμείνουμε σε επαφή και πως θα συζητήσουμε ακόμα πολλές φορές πριν την ε, κύρωση της συμφωνίας ε, ΣΕΤΑΛΑ και θα είμαστε σε επαφή και θα συνεργαστούμε στενά και για άλλες συμφωνίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Dann Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, το σημείο 10, το οποίο αφορά την λειτουργία και διαχείριση των τελωνίων ως εργαλείο για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου. Στις 25 του μήνα, την Τετάρτη δηλαδή, θα γίνει ένα εργαστήριο και θα ήθελα να παρακαλέσω να είστε όσο το δυνατόν περισσότεροι σε αυτό το εργαστήριο. Ε, παρακαλώ, όσοι θέλουν να αποχωρήσουν από την αίθουσα, να το κάνουν ήσυχα. Ησυχία, παρακαλώ. Θα γίνει λοιπόν, συνεχίζω, ένα εργαστήριο πάνω στο θέμα του πώς θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη διαχείριση στο ε, εμπόριο, στο εξωτερικό εμπόριο. Θα έχουμε πολλούς... Ε, έγκριτους προσκεκλημένους και παρακαλώ λοιπόν τις πολιτικές ομάδες να φροντίσουν έτσι ώστε τα μέλη τους να είναι παρόντα. Τώρα, υπάρχει μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, η συγγήτρια είναι η κυρία Μπεγκίν και θα της δώσω αμέσω το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, πιστεύω πως ο απότερο σκοπός αυτής της συνεδρίασής μας είναι της, ε, να, να κατανέμεται δίκαια η ευημερία και ο πλούτος. Και η ανάπτυξη, αν πιστεύουμε ότι περνά και από το εμπόριο, είναι απαραίτητο οι δικαιούχοι του εμπορίου ε, να είναι αυτοί στους οποίους στάνει το όφελος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Ο κατακαιρματισμός των τελωνιακών υπηρεσιών στην Ευρώπη οδηγεί σε τον κατακαιρματισμό των εμπορικών ροών εντός της Ένωσης. Δηλαδή, τα ευρωπαϊκά λιμάνια κάνουν ανταγωνισμό μεταξύ τους για να προσελκύσουν εμπορεύματα, όχι μόνο με βάση την αποδοτικότητά τους και την αποτελεσματικότητά τους, πράγμα το οποίο είναι θεμητό επί τη βάση των επιδόσεών τους, αλλά και ε, εκμεταλλευόμενοι τα ελλείψεις και τις διαφορές τις νομοθετικές ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Εγώ προσωπικά αποφάσισα να εξετάσω αυτό το φαινόμενο και να ανακάλυψα πόσο σοβαρό είναι. Μίλησα με πολλούς ε, ελεγκτές, ε, εκτελωνιστές που μου έδειξαν τελωνιακές εκθέσεις, οι αναφορές που ήταν λυπείς ή που δεν είχαν γίνει στην πραγματικότητα ποτέ. Αυτό επηρεάζει την εσωτερική κυκλοφορία των εμπορευμάτων και τους γιατί τα εμπορέματα πάντοτε ακολουθούν την πορεία εκείνων των χωρών όπου οι ελεγκτές είναι πιο ανεκτικοί δεν πρόκειται μόνο για την Ευρώπη, αλλά πολλές φορές ε, πρόκειται για αντικανονικότητες που διαπράττονται ώστε να προσελκυθούν οι εμπορικέ ροές προς συγκεκριμένα μέρη. Εάν η τελωνιακή πολιτική θέλουμε να είναι εκείνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να μένει ο απλός θεατής. Πολλά λιμάνια λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Και αν μιλήσουμε για τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ, θα πούνε πάντα πω χρειάζονται τεράστιε υποδομέ, περισσότερε διασυνδέσει, περισσότερε δαπάνε. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να εκμεταλλευτούμε τι δυνατότητέ μα και τα όσα έχουμε στη διάθεσή μα. Η, Ευρω... Ένωση δεν χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή πλήρω. Γι' αυτό καλώ την Κομισιόν σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσει όσο γίνεται περισσότερα τι δυνατότητε που προσφέρει η πληροφορική για να καταπολεμηθούν τα πλαστά προϊόντα και να γίνει είναι πραγματικό έλεγχο στις τελωνιακέ πρακτικές για να εμβαθύνουμε μάλλον στην ε, ε, χρήση των δυνατοτήτων όλων αυτών και στις παρακάμψεις που κάνουν τα ευρωπαϊκά, οι ευρωπαϊκά, τα ευρωπαϊκά τελώνια. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να διευκολύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να απλοποιήσουν ε, δηλαδή τις ε, τελωνιακές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα να ελέγξουν το νόμιμο εμπόριο ώστε να μπορέσουν να πατάξουν το παράνομο εμπόριο, ειδικά όσον αφορά τις εξωτερικές, ε, τις εξαγωγές μάλλον και τις εισαγωγές για να προστατευτούν οι δικοί μας έμποροι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω της, των πλαστών προϊόντων, πράγμα το οποίο θέτει σε κίνδυνο ε, πολλές θέσεις εργασίας. Έκανα τη δουλειά αυτή σε κεντρικά λιμάνια της Ιταλίας και της Ευρώπης και έχω κατανοήσει πως πολλές νομοθεσίες δεν χρησιμοποιούνται και πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες για εναρμόνιση. Ναι. Αλλά αυτή η κατάσταση βολεύει ορισμένους και γι' αυτό, όπως και στον οικονομικό τομέα, θα πρέπει να κατανοήσουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το μέρος όπου οι ισχυρότεροι γράφουν τους κανόνες και οι υπόλοιποι κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά είναι ένα σύστημα συντονισμού και συνεργασία που μπορούν, να αποδώσουν τεράστια πλονεκτήματα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο στους Κιώδης, τον κύριο Μπέντ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέντσεν. Θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια. Ε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η έκθεση που έχει προετοιμάσει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε κυρίω με αυτή την έκθεση πώ μπορούμε να απλοποιήσουμε την ε, νομοθεσία, να την κάνουμε πιο φιλική προ τον χρήστη, αν θέλετε. Και κυρίω για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Και πιο εύκολο για τη διοίκηση να την εφαρμόσει. Πάντοτε λέμε ότι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως, η Τελωνιακή Ένωση έχει δημιουργήσει πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα σε ακριβώς αυτές τις επιχειρήσεις, κάτι το οποίο δεν επιτρέπει για τη δημιουργία θέσεων εργασία. Ένα ακόμα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι τομείς στους οποίους οι τελωνιακοί έλεγχοι έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς και τους το, τομείς τους οποίους τελικά δραστηριοποιούνται εκείνοι που θέλουν να εξαπατήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες να ε, ρίξουν στην αγορά προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν η νομοθεσία πρέπει να είναι απλή, σαφής, ξεκάθαρη και για να συμβεί αυτό πρέπει να εξυγχρονιστεί η νομοθεσία περί Τολωνιακής Ένωσης. Οι προσπάθειες εξυγχρονισμού που έγιναν μέχρι τώρα δεν οδήγησαν σε απλοποίηση. Κάτι ακόμα. Για τα πληροφοριακά συστήματα προβλέπεται ε, μια μεταβατική περίοδος που λύγει το 2020. Μέχρι τότε όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν θέσεις εφαρμογή τα πληροφοριακά του συστήματα για το, την παρακολούθηση των τελωνίων. Θα ήθελα αυτό το σημείο της έκθεσης να ενισχυθεί, να γίνει πιο ξεκάθαρο, γιατί είναι ένα τομέα στον οποίο παρατηρούνται πολλά προβλήματα. Η διοίκηση στα διάφορα κράτη-μέλη δεν έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσει και δεν παρέχει τα στατιστικά στοιχεία που χρειάζονται. Η προσπάθεια εναρμόνισης της θελωνιακής νομοθεσίας πρέπει να οδηγήσει και σε εναρμόνιση των στατιστικών στοιχείων που συλλέγονται, αλλά αυτό πρέπει να οδηγήσει και σε ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας. Πρέπει επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των τελωνίων αφενός και άλλων αρχών όπως η αστυνομία ή οι κτηνιατροί ελεγκτές. Με στόχο τελικά μέσω αυτής της συνεργασίας και των συνεργειών να μειωθεί ε, η γραφειοκρατία. είναι τομεί αυτοί όλοι ε, στου οποίου πρέπει να εντείνουμε τι προσπάθειέ μα. Χαίρομαι που η συγγήτρια ε, αναφέρει την, στην έκθεση της τη σημασία που έχει διάφοροι ενδιαφερόμενοι, οι διάφοροι εμπορευόμενοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την αλυσίδα, να έχουν την ίδια ερμηνεία και την ίδια αντίληψη για την ερμηνεία της νομοθεσίας και τους κανόνες. Εάν δεν υπάρχει μια ομοιομόρφη ερμηνεία της νομοθεσίας τελικά οδηγούμαστε στις καταστάσεις ανταγωνισμού μεταξύ των, του ενός του άλλου λιμένα στην Ένωση. Θα φέρω ένα παράδειγμα του τομέα της πνευματικής ε, ιδιοκτησίας, όπου έχουμε ήδη νομοθεσία που ξεκαθαρίζει ε, ποιος είναι ο ρόλος των τελωνιακών αρχών και αυτό έχει οδηγήσει σε επιτυχίες ε, στην καταπολέμηση των ε, παράνομων αντιγράφων προϊόντων. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη νομοθεσία, αλλά καλύτερη εφαρμογή της φυστάμενης. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε κυρία Ροντρίγκες. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την ησυχήτρια ε, είναι εξαιρετική η εργασία της και πολύ καλή βάση για να αρχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το σοβαρό θέμα. Συμφωνώ με την ε, εισηγήτρια πως πρόκειται για προτεραιότητα όσον αφορά την ταχεία εφαρμογή ενός κώδικα σε ολόκληρη την Ένωση που επιτρέπει να εμβαθύνουμε ε, και να εφαρμόσουμε τις ίδιες έννοιες, να έχουμε μεγαλύτερο συντονισμό και συνεργασία ανάμεσα στις ε, αρχές. Επίσης πιστεύω ότι σε αυτό είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που έχει να παίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευκολύνει την, ε, την ε, κατάσταση, να συγκεντρώσει τις καλύτερες, καλύτερες πρακτικές και να συγκεντρώσει τα στοιχεία. Ε, ωστόσο πιστεύω πως ε, θα πρέπει να τονίσουμε κάτι ακόμα και θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες. Αυτό είναι η εναρμόνιση των ελέγχων και των επιθεωρήσεων από πλευράς των ε, τελωνιακών αρχών. Όλοι παρατηρούμε μια κατάσταση που μάλιστα έχει αναφερθεί και από το ελεγκτικό συνέδριο στην ετήσια του έκθεση όσον αφορά το γεγονός ότι το, μια ίδια διάταξη που μεταφέρεται και που εφαρμόζεται ωστόσο με διαφορετικά κριτήρια της φάση της, ε, του ελέγχου ε, οδηγεί σε παρακάμψεις της ε, κυκλοφορίας και του, των εμπορικών ροών με αρνητικό αντίκτυπο περιβαλλοντικό, οικονομικό αύξηση των καθημερινών οδικών μεταφορών ώστε να μπορέσουμε να μπορέσουν μάλλον να βρουν το πιο χαλαρό λιμάνι και τις καλύτερες συνθήκες. Εγώ πιστεύω λοιπόν πως ε, οποιαδήποτε τελωνιακή ένωση αν δεν συνοδεύεται από μια πραγματική εναρμόνιση που ελέγχει την τήρηση των κανόνων και που υπάρχουν οργανισμοί ελέγχου και επιθεωρήσεων δεν εξυπηρετεί τίποτα. Άρα λοιπόν θα ήταν καλό να δημιουργηθεί μια επιτροπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, που θα οδηγεί, θα, θα εκδίδει ε, κατευθυντήριες γραμμές, βασικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις. Επίσης πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό ε, το να καταπολεμηθεί το παράνομο εμπόριο. Θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Να μην αναφερόμαστε μόνο στα πλαστά προϊόντα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να συλλέξουμε τις ανάγκες, τι χρειαζόμαστε για να καταπολεμήσουμε το παράνομο εμπόριο. Να καταπολεμήσουμε την επιτρομοκρατία, το ξέβλημα χρήματο, το ε, ε, εμπόριο ναρκωτικών, τα πλαστά φάρμακα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών. Με αυτό νομίζω πως πραγματικά θα απηχήσουμε τα όσα μας ζητάνε οι συμπολίτες μας που μας ζητάνε δηλαδή ε, ασφαλές εμπόριο. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών, όχι μόνο ανάμεσα στους, ε, στα τελωνία, αλλά και σε όλους τους οργανισμούς που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό να προωθήσουμε την κοινωνική ευθύνη των Ευρωπαίων ε, καταναλωτών σε σχέση με την κατανάλωση παράνομων ε, προϊόντων. Ε, τα προβλήματα που αυτό προκαλεί για την υγεία, για την ασφάλεια, για το περιβάλλον και ούτω καθεξής. Είναι απαραίτητο λοιπόν να συνεχίσουμε και να δουλεύουμε για να θεσπίσουμε στρατηγικές, για να βελτιώσουμε το προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Τέλος πιστεύω πως αυτή τη φιλοδοξία θα πρέπει να προχωρήσουμε προς τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διευκόλυνσης του Εμπορίου, όπως μάλιστα αναφέρει και το άρθρο 23 της Συμφωνίας Διευκόλυνσης του Εμπορίου του ΠΟΕ, να επεξεργαστούμε συγκεκριμένους δείκτες για να αξιολογήσουμε την τελωνιακή δραστηριότητα και πιστεύω πως όλες αυτές οι πτυχές θα πρέπει να συγκεντρωθούν στην ε, έκθεση, ώστε να τεθεί πλέον τέλος σε αυτή την κατάσταση που συνεχίζεται πολλά χρόνια και εις βάρος μας. Ευχαριστώ. And, uh, merci, merci. Um, κύριε Σκάμπελ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ECR καλωσορίζει αυτό το προσχέδιο έκθεση. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή βάση συζήτηση για το θέμα. Κυρίω καλωσορίζουμε την έκκληση που απευθύνει ο εισηγητή να συνεργαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή του νέου κώδικα ε, της Ελληνιακής Ένωσης, κυρίως στους τομείς όπου υπάρχουν συντρέχουσες αρμοδιότητες, έτσι ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις σύγκρουσης. Επίσης, καλωσορίζουμε την έκκληση που γίνεται να συνεργαστούν οι κυβερνήσεις με τον ε, ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε να δημιουργηθεί μεγαλύτερη απλοποίηση ε, τη εφαρμογή τη νομοθεσία, ταυτόχρονα εξασφαλίζοντα την ασφάλεια των προϊόντων. Θα πρέπει επίση να αντιμετωπιστούν τα κενά, τα προβλήματα που υπάρχουν στου ελεγκτικού ε, μηχανισμού στα τελωνία, να, ενισχυθούν, ε, να βοηθήσουμε μάλλον τι μικρομεσαίε επιχειρήσει για να αντιμετωπίσουν το διαχειριστικό άθος από του τελωνιακού κανόνε και επίση να συνεργαστούμε με τους εμπορικούς μας εταίρους έτσι ώστε να σταματήσει η εισρωή παράνομων προϊόντων ή παράτυπων προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης υπάρχουν όμως Δύο ζητήματα που μα ανησυχούν. Πρώτα απ' όλα η εναρμόνιση των κυρώσεων και των προστήμων σε όλα τα κράτη-μέλη είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πολλέ φορέ και ε, οι ανησυχίε τι οποίε έχει εκφράσει κατά το παρελθόν το ECR συνεχίζουν να ισχύουν. Έχουμε ζητήσει πολλέ φορέ η Κομισιόν να μα δώσει στοιχεία ε, για τον τρόπο με τον οποίο οι εγκληματικέ ομάδε προσπαθούν να επιλέξουν ε, τους, τα, τα λιμάνια ή τους διόδου από τι οποίε εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουμε λάβει τέτοια στοιχεία. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί ε, ακολουθώντας τις βέλτικες πρακτικές. Επίσης μας ανησυχεί η προώθηση του συστήματος POP για προϊόντα τα οποία δεν είναι γεωργικά. Αυτό είναι πολύ δύσκολο από τη φύση τους. Από τη φύση αυτών των προϊόντων θα είναι πολύ δύσκολο να προστατευτεί η γεωγραφική τους προέλευση και θα πρέπει να ε, σκεφτούμε ότι αν προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό, μπορεί να έχουμε πρόβλημα με τι ε, φιλόδοξε συμφωνίε διεθνού εμπορίου που προσπαθούμε να συνάψουμε. Επομένω, με αυτέ τι δύο ενστάσει, ε, γενικέ γραμμέ θα υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστούμε την, ευχαριστώ την εισηγήτρια. Συμφωνούμε με την ε, γενική φιλοσοφία που έχει στο ζήτημα της Τελωνιακής Ένωσης. Κατά την άποψή μου, για να είναι αποτελεσματική, αν είναι μάλλον αποτελεσματική η Τελωνιακή ε, Ένωση, αυτό προσπίζει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε μια Τελωνιακή Ένωση η οποία να λειτουργεί. Και άρα χρειάζεται εναρμόνιση, γιατί προφανώς αν ο καθένας κάνει του κεφαλιού του, δεν θα λειτουργεί η Ένωση. και ποτέ θα καταφέρουμε να ε, καταλήξουμε σε ένα σύστημα προστασίας ε, των εμπορικών μας συναλλαγών και της οικονομίας μας. Αυτό είναι προφανές λοιπόν. Είναι προφανές ότι χρειάζεται μεγαλύτερη εναρμόνωση στον τομέα της, της ε, νομοθεσίας στα τελωνιακά. Το πρόβλημα μας το έχουν αποδείξει οι μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κανόνων σε λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σημαίνει ε, επίσης ότι χρειάζεται και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των τελωνιακών αρχών. Το σημερινό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στα τελωνιακά θέματα δεν είναι παρκές. Πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι παντού εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες και με την ίδια αυστηρότητα. Κάτι ακόμα που το ανέφεραν και πολλοί συνάδελφοι και είναι συμπληρωματικό όλοι λέμε ότι θέλουμε η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να καταπολεμεί τα παρα... το λαθρεμπόριο. Ε, και είναι προφανώς ένας, προφανώς τομέας στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη να το κάνει και έχει την ε, αρμοδιότητα και την ευθύνη να το πράξει, αλλά δυστυχώς οι δείκτες αποδεικνύουν ότι δεν τα πηγαίνουμε καλά σε αυτόν τον καταπολέμηση. Πρέπει επίση να σκεφτούμε ποια είναι η πολιτική που ακολουθούμε έναντι, πολιτικ... έναντι κρατών ε, που δεν είναι μέλη τη Ένωσης. Έχει τεθεί το ζήτημα μια Τελωνιακή Ένωση διευρυμένης στην οποία θα συμμετέχει και η Τουρκία. Εμένα με ανησυχεί αυτό, είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτική. Ε, μιλάμε τώρα να δημιουργήσουμε μια τελωνιακή ένωση με μια χώρα η οποία δεν αποδέχεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο στο σύνολό του. Αυτό πρέπει να μα απασχολήσει, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αφού λείπει η κυρία Μινέρ, θα δώσω το λόγο στο μου Τσόλτς. Θα είμαι σύντομος, Πρόεδρε, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Θα ήθελα και εγώ λοιπόν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη συνεισφορά τη και να προσθέσω ε, στο τελευταίο σχόλιο της κυρίας Δεσσαρνέζ ότι πρέπει να δούμε πώς θα αυξήσουμε τα θετικά ωφέλη της Τελωνιακής Ένωσης σε σχέση με τις τρίτες χώρες. Δηλαδή, χρειάζεται να δούμε εκ νέου τη δική μας συνεισφορά, ιδιαίτερα ε, στο τελευταίο μέρος του πρώτου κεφαλαίου του εγγράφου εργασίας. Να δούμε δηλαδή πώς θα ενισχύσουμε τη δυνατότητα ελέγχου. Όταν συζητάμε ένα σχέδιο Marshall για την Αφρική, αυτό συνεπάγεται πως θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ένα ε, σχέδιο του τι εννοούμε έλεγχος για την ε, ροή των αγαθών. Και ε, τι γίνεται στην περίπτωση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρέπει λοιπόν να το δούμε σφαιρικά. Γι' αυτό λοιπόν θα χαρώ να συνεργαστώ με την εισηγήτρια και ελπίζω να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μπούχνερ για τους πράσινους. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης. Νομίζω πως είναι μια καλή αφετηρία. Και χαίρομαι πάνω απ' όλα επειδή έγινε η πρόταση να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες σε επίπεδο ένωσης. Ωστόσο, θεωρώ πως είναι αρκετό ε, να έχουμε μία οδηγία για το πώς θα είναι η όλη διαδικασία σχετικά με τα τελωνία. Πιστεύω πως δεν είναι αναγκαίο να ε, συσταθεί μία ξεχωριστή υπηρεσία τελωνιακού ελέγχου. Εκεί που δεν χρειάζεται οδηγία είναι στις κυρώσεις. Εδώ πιστεύω πως αρκεί να υπάρχει γραμμένο στο χαρτί το τι γίνεται σε περίπτωση κυρώσεων. Τώρα, ως προς την φορολογική πτυχή, είμαι υπέρ μιας εναρμόνισης, ακριβώς διότι τα κράτη-μέλη δεν θεωρούν μόνο τα λιμάνια πολύ σημαντικά. Υπάρχει ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επίσης, να πω πως είναι πολύ θετικό το ότι η έκθεση συμπεριλαμβάνει και κάποιες περιβαλλοντικές ε, διατάξεις. Υπάρχει πρόταση για ενίσχυση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και αυτό πιστεύω θα αποβεί πολύ ωφέλιμο ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους ελιμένες ε, και πως θα αποτραπούν ορισμένοι άλλοι από το να χαλαρώσουν τους ελέγχους ε, για οικονομικό όφελος. Και αυτοί οι έλεγχοι λοιπόν πρέπει να έχουν μια πολύ έντονη περιβαλλοντική διάσταση. Γι' αυτό λοιπόν σύμφωνα με την συγχύτρια και χαίρομαι πάρα πολύ για το σχέδιο που μας παρουσίασε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Φεράν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και μάλιστα θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να σας συγχαρώ για την επανεκλογή σας. Δύο λόγια να πω η έκθεση αυτή χρειάζεται ευσεβής πόθους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει ούτε ε, οικονομική, ούτε και κοινωνική ένωση και για την τελωνιακή ένωση ακόμα λιγότερο. Υπάρχουν σήμερα χώρες που είναι πάντοτε πιο αποτελεσματικές με ένα ενοποιημένο σύστημα κοινοτικοποιημένο πολλές χώρες επιθυμούν να έχουν τους δικούς τους ελέγχους ε, για φυτο ελέγχους κυρίως και πιστεύω πως το τελωνία θα πρέπει να παραμείνουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών. Μάλιστα το διαπιστώσαμε στους τελευταίους μήνες στην καταπολέμηση της τροκρομοκρατίας υπήρξε ανάκαμψη της τελωνιακής δραστηριότητας και διαπιστώσαμε και πάλι τον απαραίτητο χαρακτήρα των τελωνιακών αρχών. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομη. Θα κάνω μια παρατήρηση. Πιστεύω πως υπάρχει μια ξενόμενη ανάγκη να εργαστούμε για πρόσβαση στις πληροφορίες όσον αφορά τις παγκόσμιες ε, αλυσίδες ε, δορυφόρων ε, ε, παγκόσμιες αλυσίδες παροχής ε, ανεφοδιασμού και βεβαίως τα τελωνία είναι πολύ σημαντικά σε αυτή την υπόθεση για όσους θέλουν να ξεκριβώσουν την προέλευση των προϊόντων. Θα πρέπει αυτό να το αναφέρουμε στην έκθεση της κυρίας Βεγγίν πιστεύω, οπότε μάλλον θα καταθέσουμε σχετική τροπολογία. Ευχαριστώ πολύ και τώρα η Επιτροπή. ποιο είναι εδώ, παρακαλώ. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, Κυρία Εισηγήτρια, αξιότιμη Κυρία Εισηγήτρια, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ που τονίζετε στην έκθεσή σας ε, την απόδοση των, τελωνίων. Η Τελωνιακή μας Ένωση εδώ και 50 χρόνια έχει δείξει εξωσημείωτη ε, ικανότητα να παραμείνει στέρεο, στέρεο θεμέλιο της Ένωσης και να προσαρμοστεί στις αλλαγές της Ένωσης και στο περιβάλλον της. Αυτό δεν γίνεται χωρίς δυσκολίες, ε, όπως τονίζεται σωστά και στο σχέδιο ψηφίσματος. Ε, εξασφάλιση της σωστής συνεργασίας ε, της, της λειτουργίας μάλλον της Ελληνικής Ένωσης χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση και διαρκής προσπάθεια ώστε να αντιμετωπίσουμε τις αναπτυσσόμενες απειλές όπως αυτές στην ασφάλειά μας καθώς και τους νέους εμπορικούς εταίρους όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο οι θεσμοί της Ένωσης και τα κατημέλη θα πρέπει να συνεχίσουν την εξέβρεση και την αναζήτηση νέων τρόπων για την αντιμετώπιση αυτών των νέων προκλήσεων. Στα διεθνή πτυχή, το γεγονός ότι η Ένωση είναι επίσης μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνίων, αυτό ενισχύει τον χαρακτήρα της Ένωσης και όπως τονίζεται στο σχέδιο ψηφίσματος, αυτό και μόνο θα πρέπει να μπορεί να επιτρέπει στην Ένωση να μιλάμε μια φωνή για τα τελωνιακά ζητήματα και να είναι αξιόπιστη απέναντι στους εμπορικούς της εταίρους σε διμερές και πολυμερές επίπεδο. Γενικότερη τώρα πτυχή η Κομισιόν πρόσφατα εκπώνησε το Δεκέμβριο ένα ανακοινοθέν για την ανάπτυξη της Τελωνιακής Ένωσης και τη διακυβέρνησή της. Αρκετέ στοιχεία αυτή τη ανακοίνωση αναφέρονται στα σημεία που αναφέρετε και εσεί στο σχέδιο ψηφίσματό σα. Τονίζεται η ανάγκη συνεργασία ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίση, αποτελεί αυτό προπόθεση για να εξασφαλιστεί η επιτυχή και η σωστή εφαρμογή των κοινών μα νομοθεσιών, καθώ και να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στα τελώνια και άλλε αρχέ που ενεργούν και υποδρούν στα σύνορα η πρόοδο που σημειώνεται στην εφαρμογή αυτή τη στρατηγική για την ανάπτυξη της Τελωνιακή Ένωση θα γίνει επί τη βάση της διετούς έκθεσης προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Τονίσατε την ανάγκη για ομοιόμορφη εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση των τελωνιακών μας κανόνων. Το γεγονός ότι έχουμε ένα κοινό σύνολο κανόνων ε, ε, είναι αλήθεια, αλλά υπάρχουν και άλλες νομοθεσίε. Το γεγονός ότι πρέπει αναπτύσσουμε μάλλον ευρωπαϊκά συστήματα μεταγραφής. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για να υπάρχει και ομοιόμορφη εφαρμογή. Όταν έχουμε κοινού κανόνες και κοινά συστήματα, ε, θέλεις να τους ε, μπορείς έτσι να τα εφαρμόσεις και με ομοιόμορφο τρόπο. Επιπλέον αναπτύσσουμε και διάφορες κατευθύνες γραμμές για να στηρίξουμε την ομοιόμορφη και σωστή εφαρμογή των κοινών κανόνων. Και η εμπλεκόμενοι φορείς ε, συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία στι ομάδε εργασίας που παρακολουθούν μαζί με την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Τέλος, η Κομισιόν έχει αναπτύξει μαζί με τα κράτη-μέλη ένα πρόγραμμα παρακολούθησης ε, της ομοιόμορφης και σωστής εφαρμογή της ενωτική ε, νομοθεσίας όσον αφορά τα συστήματα πληροφορική. Ορισμένοι ανέφεραν και η έκθεση αναφέρνει ότι το σύστημα που είναι απαραίτητο για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων και των διαδικασιών, ευλοποίηση, αλλά και ο έλεγχος που προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Τελωνιακό Κώδικα και τη μετάβαση αυτού θα πρέπει να γίνουν σεβαστοί. Φυσικά η Κομισιόν μαζί με τα κράτη-μέλη και με τους ενδιαφερόμενους φορείς συνεργαζόμαστε ώστε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο όπως έχει σχεδιαστεί. Ήδη από τώρα και βήμα το βήμα τα συστήματα IT αναπτύσσονται για να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος. Επίσης έγιναν αναφορές στο ίδιο τη επιλογή τελωνίων, ε, το γεγονός δηλαδή ότι ο κάθε έμπορος διαλέγει μια είσοδο της Ένωσης όπου η έλεγχη είναι πιο χαλαρή, λιγότερο αποτελεσματική. Αυτό δεν αποκλείεται. Πάντως η Κομισιόν έχει αναπτύξει μαζί με τα κράτη-μέλη μια στρατηγική για ένα πρόγραμμα δράση που εγκρίθηκαν το 2014 για την σωστή διαχείριση των τελωνίων. Και η έκθεση προόδου για την εφαρμογή αυτού δημοσιεύθηκε πέρσι τον Ιούλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει άλλη προσπάθεια για να εμποδιστεί αυτό ο κίνδυνος του να διαλέγει κανείς όπου τον βολεύει για να παρακάμψει ελέγχους. Αλλά αυτή η κοινή πλατφόρμα, αυτή η κοινή στρατηγική και όλες τα εργαλεία, τα επιχειρησιακά, τα νομικά, τα ηλεκτρονικά που, έχει στη που έχουν στη διάθεσή τους ελληνικές αρχές κινητοποιούνται ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει πλήρηση και αποτελεσματικός έλεγχος στα εξωτερικά μας σύνορα. Η ίδια φιλοσοφία και η ίδια προσέγγιση μας εμπνέει και στη διεθνή μας δράση αναφέρθηκε ε, η παράβαση και οι κυρώσεις, η και οι κυρώσεις, ξέρετε ότι έχουμε δύο προτάσεις επιτάπητος στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Μία ποινικοποίηση διαφόρων παραβάσεων, δεύτερη ε, προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και άλλη μία που αφορά τις παραβάσεις και τις κυρώσεις στα τελωνία. Και εκτιμούμε τη στήριξη του Κοινοβουλίου για αυτήν και τώρα περιμένουμε το Συμβούλιο να δώσει και τη συνέχεια σε αυτή την πρόταση. Θα πρέπει να σας πω ότι η Κομισιόν είναι απόλυτα προσιλωμένη στη συνεργασία με το Κοινοβουλίο ώστε να ε, εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα και για να σας αναφέρουμε πάντοτε την πρόοδο που θα σημειώνεται σε σχέση με τη λειτουργία της Τελωνιακής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Η aggiungere. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις συμβολές τους. Βλέπω πως ε, είμαστε σε, στο σωστό δρόμο για μια δεργασία που υπάρχει σύμπνοια. Η στόχη είναι κοινή. Οπότε ας προχωρήσουμε σε αυτήν την λαμπρή πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι Δευτέρα Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Εδώ λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος του σημείου 10 και θα περάσουμε αμέσω στο σημείο 11. Οι σχέσεις με την Κούβα, συμφωνία με την Κούβα, θα δώσω αμέσω το λόγο στον κύριο Μπόγκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ε, και συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Ε, προτού αρχίσω έχω κάποια σχόλια σχετικά με τη συμφωνία με την Κούβα. Δυστυχώ άρχισα να έρθω λίγο σήμερα, γιατί σήμερα το πρωί επισκέφθηκα την εκλογική μου περιφέρεια και μάλιστα με περικύκλωσαν τα πλακάτ και οι διαδηλωτέ. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Ε, πραγματικά. Είναι απίστευτο το πώς μπορούν να αλλάξουν τα γεγονότα, το πώς μπορούν να κατρακυλήσουν, αν θέλετε, ορισμένες ε, συνθήκες. Υπάρχουν ορισμένα κεφάλαια τα οποία ε, είναι καλά, τα οποία προσέξαμε την κάθε λεπτομέρεια και αυτά τα σημεία μάλιστα υποστηρίχθηκαν και από όλες τις πολιτικές ομάδες. Όμως, από την άλλη, θα είμαστε υποστηρικτές, κάτι που αρκετοί ονομάζουν ε, κίνδυνο για τη δημοκρατία. Εδώ πιστεύω πως έχουμε χάσει λίγο τον έλεγχο και πρέπει αυτοί οι λαϊκιστές να δουν λίγο πιο προσεκτικά τι σημαίνει δημοκρατία, τι σημαίνει ανθρώπινα δικαιώματα και ποια είναι τα σοβαρά πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα. Αυτά έτσι πριν αρχίσω να παρουσιάζω την έκθεση. Και θα ήθελα να το πω προτού περάσω στη συνέχεια. Τώρα, στην ομάδα παρακολούθησης, στην οποία ήμουν πρόεδρος, ε, συζητήσαμε και την Κούβα. Τους ε, τελευταίους μήνες συναντηθήκαμε και με, με τον πρεσβευτή της Κούβας. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Όμως μετά από αυτές τις συζητήσεις κατέστη σαφές πόσο μακρινός και μεγάλος είναι ο δρόμος για αυτήν την προσέγγιση. Και να πω επίσης ότι πριν από μερικές εβδομάδες είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον κάτοχο του φετινού βραβείου Ζαχάροφ, ε, εκπρόσωπο της, ε, των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Συναντήθηκα επίση με διάφορους εκπροσώπου μη κυβερνητικών οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μου επέστησαν την προσοχή στου κινδύνους που ε, ε, αντιμετωπίζουμε. Και πιστεύω πως αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μην ξεχνούμε ποτέ. Τώρα, σίγουρα κανείς δεν ξέρει τι θα φέρει η νέα κυβέρνηση Τραμπ πώς θα αλλάξει το σκηνικό στις σχέσεις των ΗΠΑ και της Κούβας. Δεν ξέρουμε ε, αν θα ε, αρθεί το εμπάργκο. Όμως ε, γνωρίζουμε ότι αυτόν τον μήνα που πέρασε ο πρόεδρος Ομπάμα ή πέρασε μία νέα νομοθεσία, το wet food, dry food, σε σχέση με τους πρόσφυγες που φτάνουν από την Κούβα στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και για πρώτη φορά οι Ηνωμένε Πολιτείε έλαβαν ε, προϊόντα τα οποία ε, έφτασαν από την Κούβα. Για πρώτη φορά η Κούβα έκανε εξαγωγές εκεί. Τώρα, αυτό που μας αφορά εδώ στην Ευρώπη είναι οι συνέπειες που θα έρθουν από την χρηματοδότηση διαφόρων έργων στην Κούβα. Το τι θα αλλάξει μετά την ε, κυβέρνηση Τραμπ. Και αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο πολιτικός ε, διάλογος, η Συμφωνία Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας με την Κούβα υπεγράφει από τους υποργούς Εξωτερικών από την ύπατη εκπρόσωπο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τον ε, Μπρούνο Παρέγια, τον Υπουργό Εξωτερικών της Κούβας. Πρέπει να πω ότι στο προσκήνιο ήταν ο πολιτικός διάλογος. Είναι εξίσου όμως σημαντικές και οι άλλες πτυχές της συμφωνίας και δεν πρέπει να παραβλέπονται. Πιστεύω πως αυτή η συμφωνία θα βοηθήσει θα ρίξει φως σε ορισμένα ζητήματα. Για παράδειγμα, θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τον πολιτικό διάλογο, τις διμερείς ε, σχέσεις και συνεργασία και θα δώσουμε ένα βήμα διαλόγου. Αλλά όχι μόνο αυτά, μέχρι και σημεία του προϋπολογισμού θα μας απασχολήσουν μετά την ε, σύναψη αυτής της συμφωνίας. Τώρα, να σας πω πως έχουμε με δώσει την σύμφωνη γνώμη μας. Από την άλλη, ζητήσαμε και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης να συνεισφέρει. Η Επίτροπος κυρία Μάλιμστρομ όπως και στην Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Κορέα, με την Κολομβία, το Περού και με τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεντρικής Αμερικής, μας ενημέρωσε σχετικά με την προσωρινή ισχύ και μας ενημέρωσε επίσης σχετικά με το ε, τι επιθυμούν. Και πιστεύω ότι παρά το ότι έχουμε μια συμφωνία μπροστά μας, πρέπει να περιμένουμε να δούμε και πώς θα τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Τώρα, θα πρέπει να συζητήσουμε και την έκθεση της ΕΕΔ. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, πώς θα συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα, αλλά να αναφερθώ σε τρία σημεία τα οποία πιστεύω πως θα πρέπει να θεωρήσουμε πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτον, ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό το αναφέρω ακριβώς επειδή από τη μία είναι ένα πάρα πολύ λεπτό και δύσκολο ζήτημα, από την άλλη όμως όταν ε, ακούω από τους διάφορους οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ε, τον ε, Φαρίνια, στον κάτοχο του ε, βραβείου Ζαχάροφ, ότι δεν μπορούσε να συναντηθεί με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν του εδόθη η δυνατότητα. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τι κρύβεται από πίσω και πώς αυτό θα καθορίσει το μέλλον. Διαφορετικά, αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, πρέπει να συζητήσουμε ίσω το ύψο του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. σω αυτό μα δώσει κάποια λύση. Μετά, έχουμε κάποια κίνητρα, τα οποία κίνητρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να ακολουθήσουμε μία γραμμή που θα ακολουθήσουμε σε σχέση με, τις, ε, με τη στάση μας για παράδειγμα, να δούμε πώς θα σταθούμε απέναντι στην επικείμενη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκμενιστάν, η οποία είναι η μόνη νευραλγική περιοχή σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε, καθώς επίσης και τα ε, εργατικά δικαιώματα, τις ε, διατάξεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης εργασίας. Ε, τώρα, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πολύ να εμβαθύνω σε αυτό, αλλά θα περιοριστώ στο να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ε, ερευνητική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χάρη στην οποία κατάφερα να δουλέψω με τον τρόπο που δούλεψα. Υπάρχει ένα ε, πρόγραμμα ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για διάφορες υποστηρικτικές ενέργειες στην Κούβα, για εξυγχρονισμό, για παράδειγμα, ε, πολλών τομέων της γεωργίας κτλ. Και νομίζω πως το Μάρτιο η κυρία Μογκερίνη είπε ότι όλοι οι φορείς της Κούβας θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτήν την χρηματοδότηση. Ας πάρουμε τον γεωργικό τομέα, για παράδειγμα. Το 21% της ε, καλλιεργήσιμης γης της Κούβας ε, το διαχειρίζεται το 54% των αγρατών. Εδώ πρέπει να φροντίσουμε για την συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα, για ένα άνοιγμα δηλαδή, έτσι ώστε να μπορούν όσο το δυνατόν περισσότεροι να υποφεληθούν από αυτές τις ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κούβα. Επίσης να πω πως με χαρά μου θα ακούσω τις προτάσεις των συναδέλφων έτσι ώστε να με βοηθήσουν στην δουλειά μου στην κατάρτιση της ε, γνωμοδότησης αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ροντρίγκε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να σας πω ότι μιλώ εξ ονόματος ε, του Σέρχιο Γκουτιέρες που είναι ο σκιώδης ζητητής και για ε, σήμερα δεν μπορούσε να είναι εδώ. Γι' αυτό μου ζήτησε εγώ να ε, σας διαβεβάσω τις απόψεις τους. Θα ήθελα καταρχάς να τονίσω ότι Αντιλαμβανόμαστε αυτή την συμφωνία ως μια ιστορική σημασία συμφωνία που ανοίγει το δρόμο στην εμπιστοσύνη στην αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κούβα ξεκινά δηλαδή μια νέα εποχή γιατί τα όσα είχαμε κάνει μέχρι τώρα ήταν απόλυτη καταστροφή. Η κοινή θέση δεν επέτυχε κανέναν από τους στόχους που ανέφερε και μάλιστα αποτελεί έναν τρόπο για να αντιλαμβανόμαστε τις πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές ε, σχέσεις που περισσότερο ανήκουν στον ε, ψυχρό πόλεμο παρά στον 21ο αιώνα. Μια τέτοια σφίση συμφωνία που είναι πιστεύω ισορροπημένη και βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στον αμοιβαίο σεβασμό και στον βασικό ρόλο που μπορεί, οφείλει και πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει τον εκδημοκρατισμό της Κούβας όπως το θέλει ο λαός της Κούβα. Και όπως είπα είναι πιο απαραίτητο από ποτέ γιατί όπως έλεγε και ο εισηγητής πρόκειται για μια αβεβαιότητα ε, το τι θα κάνει ο Τραμπ. Αυτό που είναι βέβαιο είναι τα όσα είπε στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Αυτό είναι απειλή. Αυτό δεν είναι αβεβαιότητα, είναι μια απειλή και πιστεύω πως πρέπει τώρα περισσότερο από ποτέ να προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο γίνεται πιο σύντομα να συνάψουμε αυτή τη συμφωνία, ε, να την στηρίξουμε εδώ σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο ώστε να δώσουμε μια ευκαιρία στον ε, κουβανικό λαό που μας το ζητά εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα και από την στρατηγική και γεωπολιτική άποψη η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να υψώσει τη φωνή της, ε, τη δυνατή και ενωμένη φωνή της, ε, έτσι ώστε να δείξει πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο στον οποίο θέλουμε να ζήσουμε σε σχέση με τον κόσμο τον οποίο ε, μας ζωγραφίζει ο Ντόναλτ Τραμπ. Είναι μια ευκαιρία γιατί έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε να γίνει Κούβα μέσω αυτού του, της διαδικασίας μεταρρύθμισης και οικονομικής αλλαγής. Να θεσπίσουμε λοιπόν σχέσεις βασικές πρόκειται για τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε για τον κουβανικό λαό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ζαραντήλ. Θα είμαι σύντομο. μιας και δεν έχει φτάσει το, το πλήρες τελικό κείμενο στην Επιτροπή μας. Όλοι γνωρίζουν και είχε αναφερθεί ότι μπορούμε να αναμένουμε σημαντικές αλλαγές στην Κούβα μετά τον, την εποχή μετά το Ραουλ Κάστρο που επίσης θα συνοδευτούν από σημαντικές αλλαγές στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Κούβας. Η κυβέρνηση Ομπάμα απεκατέστησε τις διπλωματικές σχέσεις και τερμάτισε το μακροχρόνιο εμπάργκο που είχε επιβληθεί ε, από τη δεκαετία του 60. Συμφωνώ λοιπόν με ορισμένους από τους προλαλήσαντες που είπαν ότι είναι άγνωστο εάν ο Ντόναλτ Τραμπ και η κυβέρνησή του θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική, θα συνεχίσει την ίδια πολιτική. Επομένως, θα ήταν σκόπιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψει το κενό και να προσπαθήσει να ε, αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο. Η θέση του ECR ήταν πάντοτε υπέρ μιας δικαιότερης και περισσότερο ισότιμης σχέσης με όλους τους εταίρους μας. Ποτέ δεν είμαστε υπέρ της λεγόμενης πολιτικής των προϋποθέσεων. Εμείς επιθυμούμε μια επικοδομητική συνεργασία. Είτε αυτό αφορά τις σχέσεις μας και τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με το Βιετνάμ, που είναι μια χώρα η οποία σίγουρα δεν έχει θετικό ιστορικό όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ίδιο υποστηρίζουμε και στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες όπως το Περού ή την Κολομβία, όταν συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση οι συμφωνίες εμπορικές με αυτές τις χώρες, εμείς πάντοτε είχαμε την κολομβια οταν συναπτει η ευρωπαικη ενωση στις συμφωνιες εμπορικες με στάση και την ίδια στάση θα προωθήσουμε και στο θέμα της Κούβας. Δηλαδή, θα επιθυμούσαμε όχι απλώς να αναπτυχθούν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με αξιωματούχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να ενισχύσουμε και το δημοκρατικό κίνημα και την κοινωνία των πολιτών στη χώρα αυτή. Σε γενικέ γραμμέ μπορώ να πω ότι αυτό είναι ένα καλό ε, σημείο κίνηση και βεβαίω θα συνεργαστούμε για τη συζήτηση αυτή. για την ΚΟΕ. Θα μιλήσω εκ μέρους του συναδέλφου Φορέντσο, ο οποίος δεν μπορεί να έρθει σήμερα. Να συμφωνήσω με όλους τους συναδέλφους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κούβα υπέγραψαν μια ιστορική συμφωνία. Και αυτό θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη σχέση ανάμεσα στα δύο μέρη. Πιστεύω πως είχαμε μια σταδιακή εξέλιξη από την έναρξη του επίσημου διαλόγου το 2008 μέχρι τώρα. Η Κούβα είναι η μόνη χώρα η οποία μέχρι τώρα δεν είχε κάποια συμφωνία διαλόγου και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς χαιρετίζουμε την σύναψη συμφωνίας, διότι θεωρούμε πως υπάρχει επιτέλους μία αλλαγή και μία στροφή από αυτήν την λογική του ψυχρού πολέμου που είχε ακολουθηθεί μέχρι σήμερα. Ελπίζουμε η συμφωνία αυτή να στηριχθεί και από το Ευρωπαϊκό και από τα Εθνικά Κοινοβούλια, διότι οι προκλήσεις και το έργο μας είναι μεγάλο η υπατεκπρόσωπος εκπρόσωπος κυρία Μογκερίνη και η κυβέρνηση της Κούβας αξίζουν την ε, συγχαρητήρια για το ότι προσπαθούν να βελτιώσουν τις σχέσεις, προσπαθούν να βρουν κοινού δρόμους. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζουμε η εκλογή Τραμπ να μην επηρεάσει την υλοποίηση της συμφωνίας αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι σαφέστατη και να προσπαθήσει να χαράξει τη δική της αναξάρτητη εξωτερική πολιτική για την Κούβα. Και τέλος, να αναφερθώ στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε πολιτικά, κοινωνικά, εργατικά και ανθρώπινα δικαιώματα. Και εδώ στην Κούβα βλέπουμε και θετικά και αρνητικά. Είναι μία εικόνα πολύχρωμη. Η Κούβα έχει κάνει μεγάλα βήματα στην ε, κοινωνική προστασία και έχουν σημειωθεί μεγάλες εξελίξεις ε, και στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ για τους πράσινους, η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτάσει σε ένα σημείο των σχέσεών της με την Κούβα όπου χρειάζεται εξυγχρονισμός της συμφωνίας. Γι' αυτό και η ομάδα μου είναι υπέρ της συμφωνίας αυτής, η οποία θα βελτιώσει πάρα πολύ την κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνούμε με τη γνωμοδότηση, η οποία θα βοηθήσει πιστεύω την Επιτροπή ΑΦΕΔ. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποια όρια, θα υπάρχουν κάποια σημεία σύγκρισης που θα πρέπει να επιβληθούν. Είναι σημαντικό όμως να υπάρχει συνοχή και να σας υπενθυμίσω εδώ ότι κάθε φορά που συζητούσαμε παρόμοιες συμφωνίες με την Κολομβία για παράδειγμα ή με άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου παρατηρούνταν κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων, απειλή κατά της ζωής κτλ. Το Κοινοβούλιο δεν είχε δείξει πάντα την ίδια στάση. Δεν υπήρχε λοιπόν αυτή η συνοχή. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι καλωσορίζω τη συμφωνία. Υπάρχουν όμω ορισμένες ευρωπαϊκές αξίες τι οποίες πρέπει να σεβόμαστε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Φερά. Η Κούβα δεν εκπληρώνει ε, μια σειρά πολιτικών κριτηρίων και θα, θα πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε συμφωνίε με τη χώρα αυτή, όπω το ίδιο πιστεύουμε και για την Τουρκία, για ε, την Τελωνιακή Ένωση με την Τουρκία. Ο κ. Βαλέσα, θα, πω, θα επαναλάβω κάτι που έχω πει και στο παρελθόν. Πρόκειται για μια ιστορική σημασία και ευκαιρία, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρώτα απ' όλα, για να μην θεωρηθεί μια ιστορική σημασία υποκρισία, στιγμή υποκρισία. Έχουμε διατρανώσει σε ολόκληρο τον κόσμο τι θεμελιώδε μα αξίε, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε την ευθύνη να ασπίσουμε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην Κούβα. Εάν δούμε τι συμβαίνει στη χώρα αυτή από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση αυτού του, κεφαλαίου, το η συζήτηση αυτού του κεφαλαίου, θα διαπιστώσουμε ότι αυξάνονται οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένω, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό το γεγονό. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται να κλείσουμε τα μάτια μας σε αυτή την κατάσταση. Το ερώτημα που θα πρέπει να θέσουμε, να θέτουμε γενικά, είναι αν οποιαδήποτε μας ενέργεια θα βελτιώσει την ζωή των κουβανών. Εάν η απάντηση είναι ναι, τότε μπορούμε να χαρούμε για το, την έκφαση αυτών των διαπραγματεύσεων. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε λόγω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδίω όσον αφορά την παροχή πληροφοριών και τη συνεργασία σα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρετε, ονομάζομαι Μπελούκνο και εργάζομαι για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια για τα όσα υπόθηκαν στη διάρκεια τη συζήτηση. Το πρώτο είναι ότι ότι η PCA ισχύει την ημέρα μετά από την υπογραφή ε, στο Συμβούλιο, εδώ στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή θα έπρεπε να έχει φτάσει εδώ κανονικά στις 13 Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό και με εντυπωσιάζει που δεν το έχετε το έγγραφο στη διάθεσή σας. Αυτό ήταν μια παρατήρηση που ήθελα να κάνω. Τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει είναι ότι εσείς μπορείτε να προχωρήσετε με τη δουλειά σας. Ε, κρεμεί η προσωρινή εφαρμογή που δεν έχει ακόμα ξεκινήσει γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί μια διαδικασία πριν να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ήθελα να αντιδράσω στην συμμετοχή ή στην εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών της Κούβας στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, να επιβεβαιώσω ότι τόσο η αντιπροσωπεία της ε, Ένωσης στην εμπλοκη τη κοινωνια των πολιτων τη κουβα στη διαρκεια των διαπραγματευσεων να επιβεβαιωσω οτι τοσο η αντιπροσωπεια τη ενωση στην αβανα οσο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση εδώ στι Βρυξέλλε, ήμασταν ανέκαθεν ανοιχτέ στην επαφή με την κοινωνία των πολιτών τη Κούβα. Υπάρχει και μια ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνεδριάζει τακτικά με Ε, ε, εκπροσώπους της ε, κοινωνίας των πολιτών που είναι αντίθετοι προς την κυβέρνηση, αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση. Αναγνωρίζουμε ότι είναι δύσκολη ακόμα η κατάσταση, το πλαίσιο είναι πιο δύσκολο από τις άλλες χώρες και ίσως αυτό να έχει καταστήσει αδύνατη την δημιουργία των ίδιων μηχανισμών όπως αυτούς που φτιάξαμε για άλλες διαπραγματεύσεις. Πάντως υπήρξε τακτική ενημέρωση προς την κοινωνία των πολιτών τόσο στην Αβάνα όσο και στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ. Το μήνυμα όμως που θα πρέπει να είναι σαφές και σαφέστατο ότι είναι ότι σαφής στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις διαπραγματεύσεις είναι ότι δεν υπάρχει προσωρινή εφαρμογή πριν από την επικύρωση από πλευράς του ε, κοινοβούλιο. Και αυτό το μήνυμα μπορείτε να το πάρετε μαζί σας και να το διαβάσετε σε όποιον δει. Δεν θα υπάρξει διοργανική συμφωνία χωρίς να, δεν μπορεί να σταθεί μια διοργανική διαδικασία χωρίς η διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακριβώς αυτό που είπατε ήθελα και εγώ να πω. Και βεβαίως η Κομισιόν μας έδωσε μια πολύ διπλωματική απάντηση που δείχνει επίση ότι το πλαίσιο και οι πραγματικέ διαπραγματεύσει με του εκπροσώπου των, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κινδυνεύουν, διακινδυνεύουν μάλιστα τη ζωή του την ίδια, οι επαφέ θα έπρεπε να είναι κάπω πιο εντατικέ και καλύτερε. Δεν χρειάζεται τώρα εδώ δημοσία να μπω σε λεπτομέρειε, αλλά είμαι έτοιμο να σα πω περισσότερα και για την Κομισιόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να κατανοήσει ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα και οι Υπουργοί Εξωτερικών και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης κάποιες φορές λαμβάνουν ένα σωρό αποφάσεις σε τέτοιου είδου συμφωνίε. Είναι μια διαδικασία μάθησης και ελπίζω πως θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο σωστό σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ βεβαίω, θα μείνω στο χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής ΑΦΕΤ και θα σα ενημερώσω αφού θα λάβουν την απόφασή τους. σα ευχαριστώ όλου πολύ. Σε ένα λεπτό θα συνεδριάσουν οι συντονιστέ και κλεισμένων των θυρών. Ένα λεπτό διάλειμμα.